Uh, Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη συνεδρίαση και να σας πω ότι στόχο έχω να συζητήσουμε πρώτα την ε, έκθεση του κυρίου Κόχ για την Ευρωπαϊκή Οδική Ασφάλεια. Η κυρία Σέντερ θα αργήσει λίγο. Ελπίζω να ε, δεχτείτε αυτή την τροποποίηση και να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν, εάν έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη, μπορώ να προχωρήσω στην έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ε, ελπίζω όλοι να είστε ικανοποιημένοι με τα πρακτικά. Πάρα πολύ ωραία. Πρωτού να δώσω το λόγο στον κύριο Κόχ να ε, καλωσορίσω μία ομάδα από την ε, ε, Ολλανδική και Αγγλική Επιθεώρηση Πλοίων. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις εδώ. Χωρίς πολλά πολλά λοιπόν. να κοιτάξουμε την ε, οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Η έκθεση του κυρίου Ντίτερ Κοχ. Ε, Ντίτερ, σου δίνω το λόγο. Ε, να πω μόνο ότι θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή, κατόπιν στους κοιόδης εισηγητές, κατόπιν θα μιλήσει ο κύριος Σίμονς από την ΕΟΚΕ που έχει εκπονήσει γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Ε, εισηγητής λοιπόν, σκιώδης εισηγητές και κατόπιν ο κύριος Σίμονς. Ja, vielen Dank, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής, τον κύριο Ντάνκνσον για την ευρύτατη υποστήριξη, αλλά και όλους τους συναδέλφους ε, για τις ε, τροπολογίες τους που πιστεύω ότι βελτιώνει κατά πολύ την εκθεσή μου. Έχω συστάσεις για την ψηφοφορία και βάλει κάπου αρνητικά πρόσημα, παρόλο που συμφωνώ με το περιεχόμενο για να αποφύγουμε ε, διπλές τροπολογίες και για να πω ότι πολλά από αυτά που ζητάτε έχουν μπει στις συμβαστικές μου τροπολογίες. Γι' αυτό έχω βάλει αρνητικό πρόσημο στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις συζητητές επίσης με τους οποίους συναντήθηκα επανειλημμένος και ε, έδειξαν και μεγάλο πνεύμα συμβιβασμού και προθυμία και τελικά νομίζω φτάνουμε στο μεγάλο στόχο της βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Στην έκθεσή μου πρόκειται για την ασφάλεια και όχι για θέματα οικονομικής πολιτικής ούτε περιβαλλοντικής πολιτικής. Έτσι, βεβαίως για τα έχω λάβει υπόψη, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Όσο λυπηρό και αν είναι που δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε την περασμένη φορά διότι απουσίαζα, χρόνο κερδίσαμε. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήρθα με το αυτοκίνητο επίτηδες για να μην παραμείνω σε κανένα σταθμό ή σε κανένα αεροδρόμιο αμανάτη. Έχουμε κερδίσει χρόνο λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε το περιεχόμενο και να εκπονήσουμε τροπολογίες συμβιβασμού. Νομίζω ότι έχω διασκεδάσει ανησυχίες συναδέλφων από όλες τις πολιτικές ομάδες γιατί καθίσαμε μαζί με τους δυο και κάναμε τουλάχιστον ε, προφορικές αλλαγές και ε, γλωσσικές διευκρινήσεις, τις οποίες θα επανέλθω στη συνέχεια. Για τη βασική δομή της έκθεσης πρέπει να πω ότι δεν είχαμε προβλήματα, ε, ούτε ως προς τους στόχους, όλοι συμφώνησαν. Ποια είναι η βάση. Επιστημονικά στοιχεία, τράπεζες δεδομένων και ορισμοί υψηλής αξίας διασταυρωμένων ε, για να βασίζεται εκεί την επόμενη δεκαετία μια φιλόδοξη πολιτική για την οδική ασφάλεια. Φιλόδοξη στόχη. Βασίζονται στα θανατηφόρα τροχέα που θέλουμε να μειώσουμε και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και δεν μιλώ μόνο για νεκρούς αλλά και για ε, σοβαρά τραυματίες. Θα πρέπει να συνεισφέρουν όλοι, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αλλά και τα κράτη-μέλη σε επίπεδο κρατών και ε, οι μεταφορικές εταιρείες, καθώς επίσης και η ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέχρι τον τελευταίο ενεχόμενο ε, στην υπόθεση αυτή των συγκοινωνιών και των μεταφορών. Θέλω να μπω σε κάποια θέματα που συζητήσαμε επανειλημμένα. Βασικό σημείο τριβής ήταν ο συντονιστής ασφαλείας, ε, της οδικής ασφάλειας συγκεκριμένα, είπα ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι καμιά καινούρια υπηρεσία, καμιά γραφειοκρατική δομή που θα στηθεί από την αρχή, αλλά να είναι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, μια υπηρεσία που να συντονίζει ε, τις Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικό, ε, Προστασία του Καταναλωτού, ε, Έρευνα, Ανάπτυξη, Περιβάλλον, ό,τι έχει σχέση με την οδική ασφάλεια. Να συντονίζεται λοιπόν η προσπάθεια αυτή που κάνουν ήδη σήμερα οι Γενικές Διευθύνσεις, αλλά αποσπασματικά και ξεκάρφωτα πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται σχεδιασμός, αλλά και συντονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται κάποιο να είναι συνομιλητής, να είναι ο κύριος υπεύθυνο. Γιατί πάνω από 36.000 είναι νεκροί κάθε χρόνο στην Ένωση, στους δρόμους μας, οπότε κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό πρότεινα το συντονιστή. Και προσβλέπω στη συνεργασία όλων σας. Διαβίου μάθηση για την οδική ασφάλεια, κυκλοφοριακή αγωγή. Είναι η αιτιολογική σκέψη ντε. Δεν χρειάζεται να πάει κανεί σε σχολείο οδηγών για να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα. Από την αρχή, από το σχολείο θα πρέπει να ξέρει. Ε, ακόμα και αν είναι πεζός ή αν ε, είναι ποδηλάτης ή αν είναι επιβάτης δημοσίων συγκοινωνιών. Ε, όλη μας τη ζωή χρειαζόμαστε για να μαθαίνουμε πώς κυκλοφορούμε στους δρόμους και τι η οδική ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε λάβαρο και σημαία μας. Έγιναν πολύ θερμές συζητήσεις για την αιτιολογική σκέψη ε να είναι υποχρεωτική οφθαλμολογική εξέταση. Το ξέρω ότι όταν θέλετε να πάρετε δίπλωμα οδήγησης χρειάζεται οφθαλμολογική εξέταση και ε, το θέμα είναι κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται. Κοιτάξτε, όταν ε, ε, κάνεις εξέταση οφθαλμολογική δεν κόβεσαι ε, ούτε σου παίρνει κανεί το δίπλωμα. Απλώ σου δίνουν κάποια βοηθήματα, γυαλιά για να μπορεί να οδηγεί. Αυτό το θέμα δεν θέλω να το βγάλω τελείω από την έκθεσή μου γιατί το θεωρώ σημαντικό. Ε, οι οδηγοί και οι επαγγελματίε οδηγοί έχουν ευθύνη και απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στους υπολείπου. Ένα άλλο τμήμα συμβασμού επίση προτείνω χωριστή ψηφοφορία για να ψηφίσουμε ξεχωριστά το υποχρεωτικό, αν θέλουμε να υποχρεωτική εφθαλμολογική εξέταση όχι. Ας το αποφασίσει η Επιτροπή μας, αν είναι ε, εθελοντικό για τους οδηγούς φορτηγών ή υποχρεωτικό. Τώρα, για το ενόπνευμα. Εγώ θα έλεγα το μήνυμά μας να είναι ότι όποιος πιάνει μόνη δεν θα πιάνει ποτήρι. Αλλά εγώ περιμένω και από τους επαγγελματίες ε, οδηγούς και από τους νέους οδηγούς να είναι το όριο πραγματικά μηδέν της χιλής. Τώρα ξέρω ότι κάποιος που παίρνει ε, διάφορα φάρμακα ή πίνει ένα χυμό ε, και αρχίζει αρχονική ζύμωση στο στομάχι του ή τρώει μια καραμέλα που έχει αλκοόλ, ε, μπορεί να έχει αποτέλεσμα που είναι πάνω από το μηδέν της χιλής. Εντάξει, ε, βασίστηκα σε επιστημονικές μελέτες και γιατρών και άλλων επιστημόνων και είπα ε, με σύμφωνη γνώμη αυτών να οριστεί. Πρότεινα και το λεγόμενο lock να είναι, μπαίνει στα νέα αυτοκίνητα με κάποιο περιθώριο ασφαλείας. Άλλη συζήτηση που έγινε. Η θέση στάθμευσης και Ασφαλή στάθμευση των, για τους επαγγελματίες οδηγούς. Και ποσοτικά και ποιοτικά. Να λαμβάνουμε όλα τα στοιχεία ε, υπόψη και όλες τις πτυχές. Ε, ε, όχι τη λογική, συγγνώμη. Ε, συμβιβαστική πρόταση πέ Το θέμα αυτών των ε, ε, γυλαίκων που θα πρέπει να φορούν ε, μόνο οι οδηγοί ή και όλοι οι επιβάτες, τι θα γίνει με τους ποδηλάτες, μόνο οι ποδηλάτες να φοράνε αυτό το γυλαίκο το φωσφορίζουν και κράνος, ποιοι θα πρέπει να φορούν αυτά τα γυλαίκα. Εγώ στην αρχή ήμουν υπέρ, αλλά τελικά κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ αυστηρές ρυθμίσεις και υποχρεωτικές. Ε, επιλέξαμε το παροτρύνει, ενθαρρύνει, encourage και το συζήτησα και με τους σκιώδεις ηγητές και κάνω αυτή την πρόταση και ελπίζω και οι πράσινοι να συμφωνήσουν. Γιατί και για τους ποδηλάτες και στην, και τη νύχτα και γενικά ε, καλό είναι να φορούν κάτι ε, που να προειδοποιεί φωτοσημαντήρε, ονομάζεται αυτό ή σήματα, δεν ξέρω κάτι που να αντανακλά το φως και να τους βλέπουν. Και ένα τελευταίο, ένα αίτημα που συζητήσαμε και συμφωνήσαμε με όλους τους συντονιστές και τους οδηγητέ χρόνια ανάπαυσης για επαγγελματίε ε, οδηγούς φορτηγών που μένουν μέσα στα φορτηγά. Και όταν κάνει ζέστη, βέβαια σήμερα δεν κάνει, ε, και δεν έχουν και κλιματισμό μέσα στο φορτηγό δεν μπορούν να αναπαυθούν. Οπότε θα πρέπει να λέμε ότι σε τέτοια φορτηγά που διανύουν μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να έχουν κλιματιστικά τα οποία να λειτουργούν ακόμα και όταν είναι σβηστός ο κινητήρας και σταθμεύει το φορτηγό. Αυτά. Περιμένω και τις απόψεις σας και με χαρά να τις ε, συμπελάβω στην έκθεσή Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I'll now go on to... Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους και εισηγητές. Αν περιοριστείτε στα πέντε λεπτά και για τους κοιόδες εισηγητές και τρία λεπτά για τους άλλους θα μπορούσαμε να τηρήσουμε το χρόνο μας. Ε, καταρχήν από τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Κόχ για την εξαιρετική δουλειά του, για το ενδιαφέρον του για το θέμα και για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων και μηνών κατά την προετοιμασία του εγγράφου αυτού. Θα ήθελα να τονίσω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια σειρά φιλόδοξων συμβιβασμών που θα μας επιτρέψουν να στείλουμε σαφές ε, μήνυμα στο ευρωπαϊκό κοινό ότι θέλουμε να ε, πετύχουμε τον φιλόδοξο στόχο μείωσης ε, του αριθμού των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων κατά 50% μέχρι το 2020. Η Σλοβενία είναι μία από τις χώρες που ήδη έχει υιοθετήσει τον στόχο μείωσης του αριθμού των θυμάτων και τα τελευταία δέκα χρόνια ε, πετύχαμε το στόχο αυτό. δυστυχώ, όμω τώρα αυξάνεται πάλι ο αριθμό των ε, τροχαίων ε, δυστυχημάτων και είναι πολλά τα, τροχαία, τα τραγικά δυστυχήματα που σημαδεύουν ολόκληρε οικογένειε. Είναι ζωτική σημασία κατά τη διάρκεια της δεκαετία αυτής να μπορέσουμε να ελέγξουμε το θέμα της υψηλής ταχύτητας και της χρήσης του αλκοόλ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους ε, συμμετέχοντες, δηλαδή τα, τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Επίσης θα ήθελα να ε, τονίσω ιδιαίτερα το θέμα της ποδηλασίας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ε, χρησιμοποιεί το ποδήλατό του, να κλείσουμε τα κέντρα των πόλεων και να περιοριστεί η κυκλοφορία εκεί σε πεζούς και ποδηλάτες. νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός ο συμβιβασμός G. τα περισσότερα ε, ατυχήματα που οδηγούν σε θάνατο ε, οφείλονται στο αλκοόλ. Γι' αυτό ε, πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή όσον αφορά το θέμα του αλκοόλ και της οδήγησης. Καθόλου η νόπνευμα λοιπόν για τους επαγγελματίες οδηγούς ε, και νομίζω θα ήθελα να καλέσω όλα τα κρατη να κάνουν ε, ό,τι μπορούν για να εφαρμόσουν το στόχο αυτό. Ήδη κάποια κράτη-μέλη το κάνουν αυτό σήμερα. Ε, είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε επιτυχία τελικά εάν αποφασίσουμε να υιοθετήσουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για τους νέους οδηγούς. Τα δύο πρώτα χρόνια με αυτό το έχουν λάβει αδειοδήγησης. Επίσης, ε, επίσης ε, να, να, χρησιμοποιηθεί το σύστημα Alcolox και ε, να γίνει υποχρεωτικό το σύστημα αυτό μέχρι το 2013. Όσον αφορά τα όρια ταχύτητας, Ε, σημαντικός αριθμός των ατυχημάτων γίνεται σε τοπικούς δρόμους ε, και είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τους πιο ε, ευάλωτους ανθρώπους. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν να περιοριστεί η ταχύτητα σε 30 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές κατοικιών και να υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι. Συμφωνώ με τη σημασία να υπάρχει χωριστή ε, ψηφοφορία σχετικά με τις ε, την εξέταση της ε, όρασης. Όσον αφορά τον, την ταχύτητα, έχουμε βρει μια πιο ήπια διατύπωση βρήκαμε συμβιβασμό όσον αφορά τη χρήση των, φωσφορι... των γυλαίκων ε, και επίσης ε, όσον αφορά την ε, χρήση τους στα αυτοκίνητα. Σίγουρα είναι ένα μέτρο που επικροτούμε. Πολύ συχνά μετά από ένα ατύχημα ο κόσμος πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο. Δεν είναι ορατή όμως διότι μόνο ο οδηγός έχει τέτοιο γυλαίκο. Επίσης, έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τον ε, ρόλο του συντονιστή. Δεν ε, ε, αποφεύγουμε την επικάλυψη εργασιών, ούτε εισάγουμε εδώ μία νέα αρχή, ένα νέο φορέα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για όλους τους συμβασμούς. Η ομάδα μου μπορεί να τους στηρίξει όλους και να, στηρίξω και να προσθέσω μία προσωπική παρατήρηση. όσον αφορά τις τροπολογίες 159 και 179. Η 159 έχει να κάνει με τα αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει ε, τα βαρέα οχήματα να μην χρησιμοποιούν ε, τα τοπικά οδικά δίχτυα όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους. Θα παρακαλούσα τον εισηγητή να επανεξετάσει ε, την ε, σύστασή του για την ψηφοφορία για το σημείο αυτό. Ελπίζω να πετύχουμε ευρεία στήριξη αύριο και επίσης όλα τα έγγραφα, όλα τα σωστά μηνύματα δεν ε, θα μπορέσουν να μειώσουν τον αριθμό των θυμάτων εάν όλες αυτές οι δεσμεύσεις δεν γίνουν πραγματικότητα και εάν τα κράτη-μέλη δεν βρουν τρόπο να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω ξανά της κυρίας Βέισβερκ γιατί ζητεί συγγνώμη, έχει ανελημμένες υποχρεώσεις και πολλές στην εκλογική της περιφέρεια και δεν μπορεί να παρευρίσκεται. Ε, ευχαριστεί επίσης τον κύριο Κοχ για τις προσπάθειες που κατέβαλε, όπως και τους υπολείπους σαν τους σκιώδης ηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων, για τη συνεργασία που ε, κάναμε και που είχαμε. Η κυρία Γκρισπέκ, λέει η κυρία Μπιλμπάου, επιμένει ότι υποστηρίζει όλες τις ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που έφτασαν μετά από μια μεγάλη συνεργασία, εκτός από τη συμβαστική β' που μιλάει για το συντονιστή και τη νέα συμβιβαστική πρόταση όπου διαφωνεί η κυρία Κρισπέκ γιατί θέλει να είναι υποχρεωτικό. Για το συμβιβασμό Β και τη δημιουργία της θέσης του συντονιστού το θεωρεί άχρηστο αυτό και πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε επιπλέον γραφειοκρατία που μπορεί να αποφευθεί και θα πρέπει να δούμε, λέει η κυρία Κρισπέκ, τι πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε. Ένα συμπίλημα, μια επισκόπηση, να δούμε ποιες πρωτοβουλίες λειτουργούν, τι δεν λειτουργεί, για να βελτιώσουμε τις ε, ισχύουσες ε, δομές. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν χρειάζεται ε, αυτός ο συντονιστής και είναι κατά της συμβαστικής πρότασης ε, Β. Σε ό,τι αφορά την ε, για το με έλεγχο τη όραση στην οφθαλμολογική εξέταση κάθε 10 χρόνια και κάθε 5 χρόνια για οδηγού άνω των 65 ετών. Συμφωνεί η κυρία Γκρίσπεκ και θεωρεί ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μέτρα που προτείνονται εδώ. Γιατί ε, η φθήνουσα όραση, η απώλεια της όρασης είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά δυστυχήματα στον δρόμο. Αλλά ε, η νέα εκδοχή του συμβιβασμού ε, δεν αναφέρει τη λέξη υποχρεωτική. Αυτό το θεωρεί σημαντικό η κυρία Γκρίσμπεκ, θέλει να ξαναμπεί. Ε, και, ε, εντάξει, να ζητηθεί ε, χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα θα υπερψηφίσει όμως τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά την ε, συμβαστική πρόταση G, ε, είχε κάποιες διαφωνίες στην αρχή, αλλά τώρα υποστηρίζει απολύτως τη νέα εκδοχή γιατί θεωρεί και καταλαβαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, απαιτήσουμε ε, μηδενική μηδενικό αποτέλεσμα ας πούμε στο αλκοτέστ είναι κάτι το ανεδαφικό. Μπορεί ένας επαγγελματίας οδηγός στην προηγουμένη ας πούμε να είχε πιει λίγο γιατί ήταν σε μια οικογενειακή γιορτή ή κάτι τέτοιο και την επομένη παραμένει στο αίμα του ο ε, αλκοολικός βαθμός και δεν είναι τελείως μηδενική εξέταση και δεν θα πρέπει αυτό να του στοιχίζει τη δυνατότητα να εργάζεται. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση του ινοπνεύματος και για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών και για τους νέους οδηγούς και νεαρούς σε ηλικία. Επίσης, ε, χαίρεται και για την προφορική τροπολογία ε, σχετικά με τον κλιματισμό στα φορτηγά αυτά, γιατί όντως θα βελτίωνε ε, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των οδηγών φορτηγών και είναι πάρα πολύ θετικό, θεωρεί η κυρία Γκρισπέκ και το υποστηρίζει. Και για τα φωσφορίζοντα γυλαίκα συμφωνεί με τις συμβεστικές προτάσεις στις οποίες κατέληξαν οι σκιώδεις Ευχαριστώ. Ο κύριο Τέλερ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ Πιστεύω πως αυτός ο αξιέπαινος ε, στόχος ε, προς ε, μηδενική, μηδενικό όραμα είναι πολύ θετική η κίνηση για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες των δρόμων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η οδήγηση δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι ένα προνόμιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να υπάρχει οδική ασφάλεια κατά λέξη δηλαδή η δρόμη να είναι ασφαλής για όλους τους χρήστες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα χήματα είναι ασφαλή και ότι οι οδηγοί τους επίσης είναι σε θέση να οδηγούν. Και καλωσορίζω τα διάφορα τεστ για την όραση και την χωριστή ψηφοφορία που είπατε για την προαιρετική υποχρεωτική φύση αυτών των τεστ. Να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί έχουμε φτάσει σε θετικό πιστεύω αποτέλεσμα εδώ. Ίσως να μην προχωράμε αρκετά όσο θέλουν κάποιοι, ίσως λιγότερο από όσο επιθυμούν άλλοι. Ε, εν περιπτώσει νομίζω πως έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο ώστε να μετατραπεί αυτή η προσδοκία για μείωση των ατυχημάτων, των θυμάτων μάλλον, ε, σε πραγματικότητα. Θέλω να εστιάσω την προσοχή σε τρεις βασικούς τομείς που ανέφεραν όλοι. Ταχύτητα, αλκοόλ και ναρκωτικά. Είμαι πολύ ε, ευτυχής που βλέπω ότι η συμβαστική φαίνεται να συνιστάται από όλα τα προς τα κρατημέλη ώστε να υιοθετήσουν ζώνες ε, ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρων στις αστικές ε, περιοχές. Και είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένο γιατί η Βρετανική κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες μόλις έκανε πρόταση ώστε η απέτηση αυτή να είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ε, τώρα για το θέμα του αλκοόλ και το αλκοολόξ και το μηδενικό ποσοστό αλκοόλ στο αίμα ήταν κάτι το οποίο είχαμε προτείνει ούτω ή άλλω, γι' αυτό είμαι ευχαριστημένο. Και όσον αφορά τα ναρκωτικά, έχουν γίνει κάποιε κινήσει ώστε να γίνεται εντοπισμό και να αποθαρρύνεται η χρήση των ναρκωτικών ε, κατά την οδήγηση. Υποστηρίζουμε την ιδέα του συντονιστή για την οδική ασφάλεια Μάλιστα, δεν πιστεύουμε πως θα υπάρχει επικάλυψη προσπαθειών εδώ, και αυτό είναι, γιατί αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θέλει να γίνει. Κανένας δεν θέλει να αυξηθεί η γραφειοκρατία, οι δαπάνες ε, και να υπάρχει επικάλυψη, αλλά δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει, γιατί με αυτόν τον συντονιστή, ε, αν γίνει έτσι όπως προβλέπετε. Τώρα, για το φωσφορίζοντα γυλαίκα, και τη χρήση τους. Ολόκληρη ιστορία, Πρόεδρε. Καταρχήν είχαμε μια έντονη σύσταση για να τα φορούν, μετά ήταν απλά σύσταση και τώρα είναι ενθάρρυνση, παρότρυνση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κρέμερ με αυτά που είπε γιατί έχει μεγάλες επαφές με τις διάφορες ομάδες δράσης των ποδηλατών και πολύ καλά μας δείχνει τις προτεραιότητες των ίδιων των ποδηλατών. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν να ευχαριστήσω και πάλι τον ε, εισηγητή. Εμείς ε, θα υποστηρίξουμε ε, την πλειοψηφία και τις συμβαστικές τροπολογίες και θα τα πούμε αύριο και στην αυρινή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπράντμπορν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να πιστέψει κανείς ότι στις παρατηρήσεις μου έχω άλλο στόχο από την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Όμως, πάντα υπάρχει ένα όμως, ένα αλλά. Κοιτάμε εδώ πράγματι θέματα τα οποία είναι απαραίτητο να νομοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι σε προηγούμενες συζητήσεις για το θέμα αυτό πάντα έλεγα ότι το ε, κλειδί εδώ είναι ε, η παλιά αγαπημένη μας επικουρικότητα. Κάποιο από τους προλαλήσαντε ε, είπε, και νομίζω ότι ε, το παραθέτω σωστά, είναι υποχρέωσή μας ως Ευρωβουλευτές ε, να αναλάβουμε δράση για το θέμα αυτό. Διαφωνώ. Δεν είναι ευθύνη μα ως Ευρωβουλευτές. Είναι ευθύνη των δημοτικών μα συμβουλίων, των εθνικών βουλευτών. Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ένωση να αναλαμβάνει δράση για το θέμα αυτό. Και αυτό είναι το σημείο εγκίνησή μου. Σε μεγάλο βαθμό, βαθμό λοιπόν ε, οι συμβιβασμοί, τα θέματα τα οποία συζητάμε μπορεί να είναι επιθυμητά, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει ε, να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φοβάμαι ότι η απάντησή μου είναι όχι. Να κοιτάξουμε κάποια παραδείγματα των συμβαστικών κειμένων που έχουμε μπροστά μας. Ε, επί πολύ καιρό συζητιέται το θέμα των χειμερινών ελαστικών για τα αυτοκίνητα. Κύριε Πρόεδρε, είναι θέμα των ε, κρατών μελών. Ήδη τα κράτη-μέλη έχουν πολιτικές, ε, τα κρατη που, το χρειάζονται έχουν πολιτική για τα χειμερινά ελαστικά. Για τα άλλα, μάλλον δεν είναι απαραίτητο να έχουν πολιτική για τα χειμερινά ελαστικά. Ας ε, μιλήσουμε για τα φωσφορίζοντα γυλαίκα. Για τον κάθε επιβάτη ε, για την μικρή πιθανότητα ότι μπορεί να ευλακούν σε ένα δυστύχημα τη νύχτα. Κύριε Πρόεδρε, θα θυμάστε ότι όταν ήσασταν νέος υπήρχε μια διαφήμιση στην αγγλική τηλεόραση, ε, στην Βρετανική τηλεόραση, που έλεγε ότι όπου υπάρχει φωτισμό τη νύχτα δεν χρειάζονται φωσφορίζοντα γυλαίκα. Α χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική. Ε, Επίση, ε, συμφωνώ απόλυτα με του φιλελεύθερου συναδέρφους όσον αφορά το επόμενο θέμα, διότι ο κίνδυνος, όπως οτιδήποτε... Ε, ε, εντός της ε, Κομισιόν ε, θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αναφέρομαι στον συντονιστή. Θα μεγαλώνει συνεχώς το γραφείο του συντονιστή. Είναι κάτι το οποίο θα μεγαλώνει όπως είναι πολύ φυσιολογικό για την Κομισιόν. Όσον αφορά τα τεστ όρασης. Γνωρίζετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πολύ καλό σύστημα ελέγχου όρασης. Τώρα λοιπόν Έχουμε ε, έλεγχο και ο οποίο επαναλαμβάνεται σε ηλικία 70 ετών. Εάν τα κράτη-μέλη θέλουν κάτι πιο αυστηρό από αυτό που έχουμε εμεί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι όμω να γίνει κάτι υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το ίδιο ισχύει όσον αφορά τα όρια για το αλκοόλ. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ε, να μην οδηγούν ε, οι μεθυσμένοι, να μην ε, οδηγούν άνθρωποι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έχουμε πολύ αυστηρή πολιτική τέτοια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν είναι απαραίτητο αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν καταδικαστείτε για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα μπορέσετε να ασφαλίσετε το όχημά σας. Η νομοθεσία λοιπόν σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν είναι πάντα ο, ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες, ε, κάποιες τροπολογίες τις οποίες μπορώ να στηρίξω. Σίγουρα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ε, οδηγούν με ασφάλεια τα ποδήλατά τους ε, με, στα σχολεία να υπάρχει σχετική εκπαίδευση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλους να έχουν κάτι τέτοιο και εννοώ το να ενθαρρύνουμε. Ε, τα κράνη στα ποδήλατα φυσικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε επίσης. Ε, ώστε να μην κινδυνεύει όποιος πέσει από το ποδηλατό του και φυσικά ε, να υπάρχουν περιοχές ε, ασφαλούς στάθμευση για τα εμπορευματικά οχήματα. Θα ήθελα κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί σε πολύ πιο ευρύ επίπεδο, διότι αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά και όσον αφορά τις ε, εγκληματικές ενέργειες ε, και, τις, ε, και τους βανδαλισμούς σε τέτοια οχήματα, το οποίο είναι πρόβλημα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για να κλείσω κύριε Πρόεδρε, λοιπόν υπάρχουν άλλοι τρόποι να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει. Όλοι θέλουμε ο κόσμο να είναι ασφαλή στο δρόμο, άσχετα από το ποιο είναι ο τρόπος ε, που μετακινούνται, ακόμα και για τους πεζούς. Ε, αυτό εδώ, όπω σα είπα, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να, ε, η νομοθεσία να γίνει στο κατάλληλο επίπεδο, δηλαδή σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σίγουρα όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, από την ΕΟΚΕ, ο κύριος Σίμων. Eh, eh. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε προχωρήσει τόσο πολύ στη διαδικασία που η δική μας συμβουλή ε, θα είναι μάλλον πενιχρή. Ε, δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, μάλλον θα έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. Πάντως, ε, αφού μας δίνετε ένα πεντάλεπτο, να σας πούμε τη γνώμη μας. Νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπόνηση της σημερινής ανακοίνωσης είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει και λαμβάνετε και εσείς υπόψη σας. Έχει σημασία το εξής γεγονός που διαπιστώνουμε. Η πρώτη στρατηγική ε, ενημέρωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από το 2000 ως το 2010 είναι πολύ σημαντική, όπως και αυτή για τη μείωση στο μισό των θανατηφόρων ατυχημάτων ή των θανάτων στον δρόμο. Αυτό είχαμε πει ήταν πολύ μεγάλη φιλοδοξία και στην επόμενη τώρα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μειώνουμε και πάλι στο μισό ε, τα θύματα από τροχέα, αλλά λέμε ότι πλέον αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη οι υπουργοί μεταφορών έχουν καταλάβει ε, πόσο σημαντικό είναι αυτό και παίρνουν και μέτρα. Αλλά όχι μόνο οι υπουργοί και ο πληθυσμός κάθε χρόνο γνωρίζει ότι θα έρθει κάποια ώρα που ο Υπουργός Μεταφορών τους θα κληθεί να ανακοινώσει τα θύματα από τροχέα στους δρόμους. Έχει γίνει λοιπόν συνείδηση η οδική ασφάλεια και στο κοινό και στον πληθυσμό και αυτό θα πρέπει να το διατηρήσουμε ως επίτευγμα και ως ε, όρμη και στόχος ε, για το 2020 είναι εφικτός. Κάναμε και μια πρόταση. Ε, να πάτε ακόμα πιο πέρα και να μην έχετε το μέσο όρο των στόχων των κρατών μελών, αλλά να διαφοροποιήσετε γιατί ξέρετε ότι ε, ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι λεγόμενες χώρες ε, sunflower και χρησιμοποιώ ακριβώς ε, τον αγγλικό όρο γιατί χρειάζομαι τα αρχικά το S, το U και το N ε, γιατί είναι η Σουηδία και ελπίζω η Σλοβενία προσεχώς, το U είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και το N είναι η Ολλανδία. Λοιπόν αυτοί οι τρεις έχουν ε, τα καλύτερα επιτεύγματα και είναι πολύ δύσκολο να μειώσουν τον αριθμό των θυμάτων στο μισό, γιατί έχουν ακριβώ τόσο λίγα θύματα, δυσκολεύονται δηλαδή από τις καλέ τους επιδόσεις. Και δεν θα πρέπει να έχουμε μία ισοπαίδωση ε, και των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες. Επίσης, και στην Επιτροπή κάναμε ε, και δώσαμε μάχη και για το ποσοστό και το δίκτυο ε, αλκοολεμίας, όχι μόνο στα φορτηγά αλλά και στα γιοταχή. Ακούω πολλά εδώ για οδηγούς φορτηγών. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τους οδηγούς ε, αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, γιατί και ε, στόχος ε, είναι και αυτή στη γνωμοδότησή μας, εντάξει όχι τόσο φιλόδοξος, αλλά απορρέει από τις συζητήσεις που έγιναν στην αρμόδια επιτροπή. Κάτι άλλο που δεν διαβάζω επίσης τόσο πολύ στην έκθεση είναι η πρότασή μας να γίνονται αιτήσιοι έλεγχοι ε, στα μαύρα σημεία της κάθε χώρας, στους εθνικούς οδικούς χάρτες, στις καρμανιόλες τις λεγόμενες ε, και στα σημεία ε, που έχουμε τα περισσότερα θύματα να γίνονται αιτήσιοι έλεγχοι. γιατί οι χώρες θα πρέπει να επενδύσουν ακριβώς για να διορθώσουν τα κακό σκήμενα σε αυτά τα σημεία που είναι τόσο επικίνδυνα. Λοιπόν, για τους στόχους, είπαμε ότι τους έχουμε διατυπώσει, μείωση των θυμάτων στο μισό, των θανάτων δηλαδή, αλλά θύματα για μας είναι και η σοβαρή ε, τραυματίες και επίσης θα πρέπει να εναρμονιστεί ο όρος ελαφρός τραυματισμός, γιατί δεν είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη. Επίσης θεωρεί η Επιτροπή ότι 25% των ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που δεν είναι ε, ενεχόμενα συνοδική ασφάλεια θα πρέπει να ενταχθούν στα 10 στα υπόλοιπα με την διαβιουμάθηση, με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση αλλά αυτά τα λένε και οι τροπολογίες σας. Κάτι άλλο που είδαμε εμείς στις εργασίες μας είναι ότι χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση για την ε, αστυνομία, την τροχέα δηλαδή, ε, την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα. Γιατί δεν γνωρίζουν πολύ καλά ε, πώς να δρούν και πώς να αντιδρούν σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις και τις τόσο σοβαρές. Και η Επιτροπή μας λοιπόν ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα και ελπίζω να σας ενημέρωσα κυρίως για τα θέματα που αναφέρονται λιγότερο στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα περάσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Παρακαλώ να περιοριστείτε στο τρίλεπτο. Ξεκινάω με τον κύριο Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κοχ για την πολλή δουλειά που έχει κάνει και για τους ε, φιλόδοξους ε, στόχους που έχει θέσει. Ε, και όσα ακούω εδώ δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα για την πολιτική μου ομάδα. Θα ήθελα να ε, συνδέσω το θέμα αυτό με το επόμενο θέμα, την ε, διασυνοριακή ε, δίωξη, διότι παρά την ευαισθητοποίηση και τα μέτρα στο, στην εκπαίδευση, πάντα θα, πάντα θα εμφανίζονται θέματα ποινική δίωξη διασυνοριακής. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει συμφωνία και για το θέμα αυτό όσον αφορά τον συντονιστή. Ε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ακόμα και αν, είμαι, ακόμα και αν προσωπικά είμαι της άποψης ότι Υπάρχουν πολλά θέματα εδώ τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, ε, να αποτελούν αντικείμενο εποπτείας και τα θέματα που αναφέρθηκαν όπως για παράδειγμα οι θέσεις στάθμευσης ε, ήδη ξεφεύγουν από το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ε, το θέμα εδώ είναι η ε, ασφάλεια των οδηγών, οπότε είναι αμέσως, αμέσως κοινωνικό το θέμα. Ε, υπάρχουν πολλά λοιπόν ε, θέματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμού πέρα από την ε, οδική ασφάλεια αυτή καθ' αυτή. Είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος, καταλαβαίνω όμως ότι η πρόταση έχει γίνει στο πνεύμα συμβασμού και θα την στηρίξω. Επίσης, νομίζω ότι όσον αφορά την ποδηλασία έχει βρεθεί καλός συμβιβασμός και Ε, όσον αφορά την ε, τροπολογία 35, ε, νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε με τα Ηνωμένα Έθνη που έχουν θέσει ένα σχέδιο για την οδική ασφάλεια. Στόχος είναι να προστατεύσουμε τους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία αλλά και τις οικογένειές τους τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Θυμάτων ε, Τροχαίων Δυστυχημάτων που είναι και παρόν. Ελπίζω οι συνάδελφοι να στηρίξουν τι προτάσει αυτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Τρία λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. <laughs> Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με τα συγχαρητήρια προς τον κύριο Κοχ για την επιμονή του και ε, την υπομονή του για να βελτιώσουμε αυτά τα θέματα της οδικής ασφαλείας και κυρίως ε, για να τα διευρύνουμε σε νέες προκλήσεις, σε νέα πεδία, γιατί ο στόχος της μείωσης των μισό των θυμάτων από τροχέα είναι πολύ σημαντικός και όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέονται και με τη μείωση των τραυματιών είναι ε, καινούρια πεδία και θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το πνευμά και τα όρια, πέρα από το γεγονός ότι συμφωνώ απολύτως με αυτή τη θεώρηση να τίνουμε στο μηδέν και να είναι ο τελικός μας στόχος για τον απόλυτο περιορισμό, Λυπάμαι που επικεντρωνόμαστε μόνο στους επαγγελματίες και δεν ε, το επεκτείνουμε και στους υπολείπους. Και μιλάμε μόνο για τους νέους οδηγούς, τους νεαρούς οδηγούς που είναι όλο και λιγότεροι γιατί είναι όλο και λιγότεροι νέοι στην Ευρώπη και δεν κοιτάμε τι γίνεται με τους ενήλικες και με τον πληθυσμό που γερνάει και δεν είναι επαγγελματίε και αρχίζουν και πειράζονται όχι μόνο από ναρκωτικά, γιατί δεν παίρνουν όλοι ναρκωτικά, αλλά παίρνουν φάρμακα όσο προχωράει η ηλικία και αυτά επιδρούν στην οδήγηση. Ε, αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να τους συμπεριλαμβάνουμε και αυτούς στον έλεγχο. Εδώ υπάρχει έλλειμμα ελέγχου, όχι μόνο επαγγελματίες λοιπόν και οι νέοι οδηγοί. Επίσης, συμφωνώ και για το συντονιστή και για την παγκόσμια ημέρα και όλα αυτά που θέλετε. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία ε, για να πετυχάνουμε τους στόχους μας, αλλά και το συμβουλευτικό φόρουμ. Επιτύχαμε και όπως και στο θέμα των διασυνοριακών παραβάσεων και Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν ε, ότι είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε στη διαβούλευση όλες τις αρχές, τις αστυνομικέ αρχές, τα θύματα, ε, ε, ε που γνωρίζουν πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες και καθημερινά μας βοηθούν για να βελτιώνουμε τη νομοθεσία μας και τα θέματά μας. Θέλω μόνο να πω για το μέλλον τονίσατε εσείς αυτό το θέμα των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπαίδευση, όντως ο στόχος, αλλά και ηλικιωμένοι ή εκείνοι που οδηγούν δίτροχα ε, με κινητήρα, μοτοσυκλέτες συγκεκριμένα, ε, ε, έχουν πολύ μεγάλες απώλειες τους αυτοκινητοδρόμους. Και σε αυτούς θα πρέπει να στραφούμε για τα αυριανά μας μέτρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σα συγχαίρουμε για τους στόχους σας και σιγά σιγά μπορούμε να συμπεριλαμβάνουμε και νέες προκλήσεις και νέες κατηγορίες χρηστών για να μειώσουμε τη... τα ατυχήματα και τα θύματα. Η κυρία Μάισνερ, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόχ. Νομίζω ότι ε, έχει εκπονήσει πολύ σοφά τους ε, συμβιβασμούς, διότι κάποιοι ε, έχουν πολύ ήπια διατύπωση. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Αναρωτιέται κανείς ε, λοιπόν σε τι βαθμό ε, χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι νομοθετική η έκθεση αυτή, είναι, πρόκειται για συστάσεις. Αναφέρεται λοιπόν η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Κυρίως ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα. Βρίσκω πολύ σοφούς του συμβασμούς σας, όπως ε, είπα ήδη, ε, όπως τον συμβασμό ε, όπου η κυρία Πιλπάου είπε εκ μέρους της κυρίας Κρίσπεκ, ότι θα γίνει χωριστή ψηφοφορία για το υποχρεωτικό τεστ. Ε, ξέρω ότι δεν συμφωνούν όλοι με την ε, κυρία Βιλπάου. Ε, έτσι λοιπόν θα μπορούν κάποιοι να υπερψηφίσουν την τροπολογία ακόμα και αν είναι κατά της, του υποχρεωτικού τεστ όρασης. Μπορεί να αναρωτηθεί κανείς ε, εάν ε, πρέπει να προχωρήσουμε στο βαθμό που αναφέρει η αρχική έκθεση, για παράδειγμα ε, τα φωσφορίζοντα γυλαίκα. Εμείς ως φιλελεύθεροι αναρωτιόμαστε σε τι βαθμό είναι απαραίτητο να λάβουμε απόφαση. Ξέρω ότι οι ποδηλάτες είναι ευάλωτοι, αλλά το να τους αναγκάσουμε να φορούν φωσφορίζοντα γυλαίκα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ακόμα και αν γαλλικοί σχεδιαστές έχουν ε, φτιάξει πολύ ωραία γυλαίκα. Επίσης, ε, όσον αφορά τον ε, συνάδελφο Κέιλερ, μπορεί κανείς να πει ότι το να διηγεί κανείς αυτοκίνητο είναι προνόμιο, ωστόσο κάποιοι πρέπει να το κάνουν αυτό λόγω του, της δουλειάς τους και νομίζω γι' αυτό μπορούμε να είμαστε κάπως πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις ε, διατάξεις. Ε, τρία θέματα ακόμα. Ε, συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά τον συμβιβασμό J, διότι αναφέρεται στην παθητική ασφάλεια που μπορεί να βελτιωθεί με περισσότερες έρευνες. Ο συμβιβασμός είναι επίσης ένας τομέας όπου μπορεί κανείς να προχωρήσει περισσότερο και η τελευταία τροπολογία αφορά τα κλιματιστικά ουσιαστικά ε, τίθεται πάλι το θέμα εάν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι είναι, σημαντικό. Ε, στα νέα φορτηγά ε, ε όντω υπάρχουν αυτέ οι εγκαταστάσει. στα παλιά μπορεί κανεί να το κάνει αυτό με χαμηλό κόστο. διότι η ξεκούραση των οδηγών φορτηγών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αν μπορούν να ξεκουραστούν μέσα σε ένα κλιματιζόμενο φορτηγό. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Φαντάλεν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κανείς δεν διαφωνεί με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ε, πατάμε γερά στη γη, όχι εθεροπάμονες. Ε, και σε αυτά που έχει πει ο κύριος Κόχ, έχει δίκιο σε πολλά σημεία. Ε, και εγώ συμφωνώ με την εναρμόνιση ε, του θέματος των ορών ανάπαυσης. Είδαμε τι σημαίνει μη εναρμόνιση, το έχουμε ζήσει και στο πετσί μας και αυτό το σχέδιο Βερόνικα είναι πολύ καλό, αλλά από την άλλη έχει και κάποια στοιχεία με τα οποία δεν συμφωνούμε. Το θέμα του συντονιστού ή τα ελαστικά, τα χειμερινά. Ε, αυτά που λέτε για τους ποδηλάτες. Εγώ κάνω πολύ ποδήλατο στη χώρα μου, έχω ποδήλατο και στο Στρασβούργο μόνιμα και εκεί κάνω ποδήλατο. Και κινδυνεύω να φάω κλίση άμα ξεχάσω το γυναίκο μου στο Στρασβούργο. Ε, νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τα άλλα δεν έχει και πολύ μεγάλες αρμοδιότητες. Εγώ θα χαιρόμουν πολύ περισσότερο ε, να έκανε και που ε, έκανε πραγματικά υποδομή για τους ποδηλάτες η τοπική αυτοδιοίκηση και φτιάχνει και ποδηλατόδρομους και μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Αυτά ωραία. Αλλά τώρα τα γυλαίκα εντάξει. Κάτι άλλο. Ε, το θέμα της φιλοδοξίας. Στην παράγραφο 7 λέει ότι θα πρέπει να κατα ε, τίνουμε προς το, ε, το μηδέν. Ε, κανένα θύμα στους δρόμους. Εντάξει, ωραίος στόχος είναι αυτός και ευγενής, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε μηδέν θύματα στον τύπο, στον δρόμο, συγγνώμη. Και να βγούμε στον τύπο και να πούμε, κοιτάξτε τι φοβερός που είμαι και συγκινητικός. Όλα αυτά μπορεί να είμαστε, αλλά δεν είμαστε και θεροβάμονες. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ποτέ κανένα νεκρό στους δρόμους μας. Νομίζω είναι υπερβολικά αυτά που γράφεται σε μερικά σημεία και αυτό σημαίνει ότι αύριο το πολύ αποχή. Ε, δεν σας το υπόσχομαι, μπορεί και να καταψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο ε, Κράμερ, τρία λεπτά. Ε, ναι, η έκθεση έχει βελτιωθεί με ε, τους συμβασμούς. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ στην συμβαστική τροπολογία για τα φωσφορίζοντα γυλαίκα. Σημαντικότερο από όλα είναι να έχουμε επιστημονικά στοιχεία. Στον συμβιβασμό αυτό έχουμε την περίπτωση ενός ατυχήματο που πρέπει να έχει φωσφορίζον γυλαίκο σε περίπτωση ατυχήματος ε, και τον εξισώνουμε με το ποδηλάτι που πρέπει κάθε μέρα ε, να φοράει ε, γυλαίκο. Δεν θα πρέπει να συνδέσουμε τις δύο αυτές περιπτώσεις. Δεύτερη περίπτωση. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι το 90% όλων των ατυχημάτων με αυτοκίνητα και ποδήλατα στις 90, στο 90% των περιπτώσεων φταίει το αυτοκίνητο. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ε, μιλάμε για ε, ε, υπερβολική ταχύτητα του αυτοκινήτου. Αυτό όμω δεν το αναφέρεται καθόλου. Δεν αναφέρεστε καθόλου στα όρια ταχυτήτων, ούτε στον αυτοκινητόδρομο, ούτε αλλού. Γιατί λοιπόν είναι τόσο επικίνδυνο, διότι ξέρουμε στις στατιστικές όπου εκεί όπου υπάρχουν πολλά ποδήλατα έχουμε τις τα λιγότερα ατυχήματα στις κάτω χώρες και ε, στη Δανία. Ε, εκεί που έχουμε τα λιγότερα ποδήλατα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ε, τα περισσότερα ατυχήματα. Αν λοιπόν θέλουμε να ε, προστατεύσουμε τους ποδηλάτες πρέπει να ενθαρρύνουμε πολλούς να πάρουν το ποδήλατό τους, έτσι θα μειωθούν τα ατυχήματα. Όταν ε, εισάγανε τα κράνη στην Αυστραλία πέσαν κατά 50% οι ποδηλάτες και αυξηθήκανε τα ατυχήματα. Όλα αυτά λοιπόν ε, δεν ταιριάζουν ε, με τις προτάσεις σας, διότι κάνετε τα θύματα ε, κατηγορούμενος. λέτε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το ποδήλατο, διότι ο ποδηλάτης είναι το θύμα και είναι ο πιο ευάλωτος. Ε, στο Η Ηνωμένο ε, ε, Βασίλειο έγινε μια δοκιμή με ποδηλάτε ε, που οδηγούσαν με ή χωρί κράνο. Όταν λοιπόν φορούσε κράνο ο ποδηλάτη, το αυτοκίνητο περνούσε με μεγαλύτερη ταχύτητα και πολύ πιο κοντά στο ποδήλατο, διότι ο οδηγό του αυτοκινήτου θεωρούσε ότι α, προστατεύεται αρκετά. Και αν πρέπει το, ο ποδηλάτη να φοράει τέτοιο γυλαίκο, γιατί να μην φοράνε κήπεζοι. Ο θα χαιρόταν στην Κίνα αν όλοι φορούσαν τέτοιο τέτοιο γυλαίκο. Και Ε, γιατί δεν λέτε αυτοί που οδηγούν καμπρίολε να φορούν Ε, αυτοί είναι ε, οι, πιο ευάλωτοι. Ε, ε, συγκεντρώνεστε μόνο στους ε, ποδηλάτες. Ε, γιατί να μην φοράνε εκεί πεζί στο σκοτάδι τέτοια γυλαίκα. Τέτοιες διατάξεις δεν επιτρέπεται να υιοθετήσουμε. Γι' αυτό είμαι κατά του συμβιβασμού αυτού και είμαι υπέρ ε, χωριστής ψηφοφορίας. η περίπτωση ατυχήματος σε αυτοκινητόδρομο που πρέπει κανείς να έχει γυλαίκο δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή ζωή ζωή ενός ποδηλάτη. Ε, ε χρειάζομαι τρία-τέσσερα γυλαίκα επειδή έχω τρία-τέσσερα ποδήλατα. Αυτή είναι λάθος οπτική. Ε, ε είμαι πεπισμένο ότι αν οδηγούσατε περισσότερο ποδήλατο δεν θα ε, σκεφτόσασταν τέτοιε. Δεν θα σα έρχονταν τέτοιε ιδέε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάικλ. Νομίζω ότι η Κίνα του ΜΑΟ θα χαρεί πάρα πολύ, διότι ε, αυτοί μάλλον θα φτιάχνουν όλα τα γυλαίκα, τα φωσφορίζοντα. Ο κύριο Χίγκιν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, και οι άλλοι ε, ομιλητές, ε, συμφωνώ με τους συμβασμούς. Πιστεύω ότι είναι πολύ ισορροπημένη η έκθεση αυτή. Στο κάτω-κάτω θέλουμε να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε τον αριθμό των θυμάτων στο δρόμο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις υποχρεωτικές διατάξεις όσον αφορά την οδική ασφάλεια και το κλειδί στο κάτω-κάτω είναι η επιβολή του νόμου. Θα πρέπει να θέσουμε κανόνες, ε, πρότυπα ε, και διατάξεις, ε, διότι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσουμε με το εγχείρημα αυτό. Αυτό που έχει κάνει εδώ ο είναι ότι έχει πάρει μια σειρά κοινών διατάξεων που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη και τις έχει βελτιώσει. Εγώ θα έλεγα εδώ ότι μένουμε στην Ευρώπη όπου έχουμε ε, ανοιχτά σύνορα ε, και υπάρχει μεγάλη κίνηση ε, οχημάτων από τη μία χώρα στην άλλη και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κοινή σειρά προτύπων και διατάξεων. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όσον αφορά τις τροπολογίες θα ήθελα να επικροτήσω μια σειρά τροπολογιών η πρώτη, ε, στην οποία, ε, η πρώτη παρατήρησή μου είναι ότι η χώρα μου έχει ε, εποφεληθεί πολύ από τα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε φτιάξει αυτοκινητοδρόμους, δυστυχώς όμως τα περισσότερα τροχιά μας θύματα δεν είναι στον αυτοκινητόδρομο και γι' αυτό επικροτώ το θέμα της βελτίωσης της ε, εποπτείας ε, στους μικρότερους δρόμους, ε, διότι δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά στη δική μου εκεί γίνεται η πλειοψηφία των ατυχημάτων. Δεύτερον, επικροτώ το γεγονός ότι ο εισηγητής έχει δεχτεί την τροπολογία μου. Είναι αποδεδειγμένο ότι Ε, όταν γράφει κανεί μήνυμα στο κινητό του, 5 στα 6 δευτερόλεπτα ε, έχει αποσπαστεί η προσοχή του, ακόμα και αν ε, είναι πολύ έμπειρος σε αυτό. Και ε, τρεις έπρεπε να φέρω στην Επιτροπή Αναφορών που έχασαν ε, τις ε, κόρες τους λόγω κακής σήμανσης στον δρόμο και γι' αυτό επικροτώ το γεγονό ότι η έκθεση ασχολείται με το θέμα αυτό και τέλο, εξίσου σημαντικό όμως, είναι το τεστ όρασης για του οδηγού. Ε, από ό,τι κατάλαβα, Εάν υπάρχει μοντέλο καλή πρακτική στη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό στι τέσσερι αυτέ χώρε, γιατί να μην ε, εφαρμοστεί στι ε, υπόλοιπε χώρε. Στο Βέλγιο δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο τεστ. Στη Γαλλία, αν μπορεί κανεί να διαβάσει μια πινακίδα οχήματο, μπορεί να πάρει αδιαδίγηση. Και τέλο, επικροτώ την τροπολογία σας ε, για, ε, τα, ε, για τις μηχανές. Θα ήθελα να σας συγχαρώ λοιπόν για, το, για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τον Τίτερ για την έκθεσή του και να κάνω τρεις παρατηρήσεις Χωρίς να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν προηγουμένως, η πρώτη παρατήρηση αφορά την επικουρικότητα. Και φυσικά βρισκόμαστε σε μια χνομοδότηση, αλλά όσο περισσότερο ανεβάζουμε τα πρότυπα, τόσο περισσότερο θα έχουμε πρόβλημα επικουρικότητας, γιατί τόσο περισσότερο θα έχουμε αντίκτυπο στις εθνικές νομοθεσίες. Όσο πιο απαιτητικοί είμαστε δηλαδή σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο θα έχουμε προβλήματα. Το ίδιο έγινε με την περιορισμό της ταχύτητας στα 30 ή στα 20 χιλιόμετρα την ώρα και εκεί ε, προσκρούμε στην εθνική επικουρικότητα. Είναι αλήθεια ό Ισχύει γενικά αυτό όταν μιλάμε για πρότυπα. Επίσης, ε, εξέταση όρασης. Θα ήθελα ως ε, γιατρός να κάνω την εξής παρατήρηση. Υπόθηκε ότι το να οδηγεί κανείς είναι ένα προνόμιο είναι και ανάγκη όμω για πολλού ανθρώπου και όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Σκέφτομαι και ανθρώπου που κατοικούν στην Ήπεθρο ή το τι αντιπροσωπεύει αυτό για τα άτομα τα πιο ηλικιωμένα για την δυνατότητα κινητικότητα. Αν βάλουμε τέτοιες, <coughs> τέτοια τεστ ε, σωματικών ικανοτήτων. Γιατί μόνο να πούμε για την όραση, ας μην ή να μην πούμε ότι μπορεί να υπάρχει αναπηρία στο κινητικού τύπου, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι τα προοδικά ε, αυτοκίνητα, γιατί έχετε κάποιο τέτοιο αναπηρία, ε, όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα σκεφτούμε, αν πάμε δηλαδή σε μια πλήρη ιατρική εξέταση. Με εντυπωσιάζει δηλαδή που σκεφτόμαστε μόνο την όραση. Άμα ξεκινήσουμε τέτοιου είδους εξετάσεις, πού θα βάλουμε το όριο. Είστε πολύ καλά, λιγότερο καλά, καθόλου καλά κτλ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πρέπει κανείς δηλαδή να είναι σε απόλυτα καλή φυσική κατάσταση για να οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει ένα κατόφλι ανοχή σε ποιο επίπεδο και για ποιο είδος προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Είμαστε βέβαια στο πλαίσιο μια γνωμοδότηση, αλλά όταν κάνουμε μια γνωμοδότηση, μην ξεχνάτε ότι δίνουμε την αίσθησή μα. Και σε κάποιε περιπτώσει αυτό μπορεί να σταματήσει το Συμβούλιο, που θα πει ότι ποτέ δεν πρόκειται να συνοηθούμε με το Κοινοβούλιο, το δούμε και σε άλλα θέματα. Οπότε α τα αφήσουμε καλύτερα. Τρίτη παρατήρηση. Λυπούμε που η τροπολογία 88, την οποία εγώ υποστήριξα, δεν γυροδεκτεί γιατί θέλει να καταστήσει το σύστημα της υποχρεωτικής ζώνης ασφαλείας Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλο, υπάρχει μεγάλος αριθμός θανάτων που οφείλεται στην ε, ζώνη ασφαλείας. Θα, οι κατασκευαστές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα να βάλουν και ένα κλείδωμα στην ζώνη ασφαλείας. Εντάξει, το μηδέν, ε, μηδέν ε, θάνατοι είναι υπερβολικό, αλλά το να υπάρχει μια ασφάλιση της ασφάλειας, της ζώνης ασφαλείας, δεν νομίζω πως είναι τόσο τρομερό και είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ, κύριε Τικάου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών, των, εθνικών αρχών, των τοπικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο βαθμό των αρμοδιοτήτων που έχουν αρμοδιότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια θα είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι, μεταφο... οδικές ε, υποδομές, δηλαδή οι δρόμοι κυρίως. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και σωστή σήμανση, σήμανση των ε, έργων στους δρόμους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συστήματα μεταφορών τα οποία να βοηθούν την μείωση των συμφορήσεων και αθώς και να ειδοποιούν σε πραγματικό χρόνο για ατυχήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα συστήματα GPS. Επίσης είναι σημαντικό να συμμετέχουμε και να βοηθούμε τους ευάλωτους χρήστες των δρόμων, όπως οι ποδηλάτες, οι πεζοί, τα παιδιά, Είμαι υπέρ της χρήσης ε, της ε, υποχρεωτικής χρήσης κράνους για τους χρήστες των δρόμων καθώς επίσης και υπέρ των ε, γυλαίκων, των φωσοριζόντων γυλαίκων. Ωστόσο, κυρίως το κράνος είναι που ωφελεί, που χρησιμεύει. Οι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει ζωή τους επειδή δεν φορούσαν κράνος. Να αναφερθώ τέλος στο μάξιμο όριο για το αλκοόλ. Θα πρέπει να επιμείνουμε για την μηδενική ανοχή. Πρόσφατα στην Γαλλία σε ένα πάρκινγκ είδα ότι μπορεί κανείς να αγοράσει αλκοοτέστ. Όποιος όμως αγοράζει ένα τέτοιο αλκοοτέστ ήδη αναρωτιέται για την ε, περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα του. Γι' αυτό και θα ήταν ε, πιο ασφαλές αν υπήρχε μηδενική ανοχή για το αλκοόλ στο τιμόνι. Ε, θα ήθελα να συνεχαρίσω τον κύριο Κοχ. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες, αλλά φτάσαμε σε καλή συμβιβαστική. Ελπίζω ε, ότι όλες αυτές οι συστάσεις θα επιβληθούν κιόλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Πιστεύω ότι έχει καταφέρει πολύ καλά ε, να αντιμετωπίσει το θέμα των ε, τροπολογιών. Όσον αφορά την ε, τροπολογία ΙΤΑ, Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση σε έξι κράτη-μέλη που ε, ισχύει η μηδενική ανοχή και να εφαρμόσουμε τα ίδια μέτρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και επίση όσον αφορά την ε, τροπολογία 141, ε, τα θύματα στους ε, μικρούς δρόμους. Ε, θα ήθελα να στηρίξω την δημιουργία πιο ασφαλούς υποδομής και σε άλλους δρόμους πέρα από τους αυτοκινητοδρόμους. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εγώ ίδιος. Ε, καταρχήν ε, να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, πολύ καλή έκθεσή του και να συγχαρώ και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους στην προσπάθεια να έχουμε μια συνεκτική έκθεση. Από τη φύση της λοιπόν η έκθεση αυτή είναι γεμάτη συμβιβασμούς. Κάποιοι θα θεωρήσουν ότι είναι υπερβολικοί, κάποιοι θα θεωρήσουν ότι δεν αρκούν. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό ότι το Κοινοβούλιο παρουσιάζει μια θέση που αφορά την οδική ασφάλεια. Δεν είναι πρώτη φορά που το έχουμε κάνει αυτό, όπως γνωρίζει ο ίδιος ο Ντίτερ. Ωστόσο, συνεχίζουμε να βλέπουμε ατυχήματα στο δρόμο σε ε, όχι πολύ καλό ποσοστό. Ε, αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να νομοθετήσουμε ώστε να αποφύγουμε την ανθρώπινη βλακεία. Διότι όταν ε, κοιτά κανείς ε, τι γίνεται στο δρόμο, εγώ συνεχίζω να βλέπω Παρότι στη χώρα μου υπάρχει σχετική νομοθεσία, βλέπω τον κόσμο να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο την ώρα που οδηγεί. Βλέπω μικρά παιδιά, μωρά, στα, στην μπροστινή θέση στο αυτοκίνητο. Μαζί με περίπου 10 ε ε, ε, ε, αστυνομικούς ε, της τροχέας. Ε, είδα τους, ε, ε, τους ηλίθιους που προσπαθούν να περάσουν ε, την, ε, τις γραμμές τη στιγμή που πλησιάζει τρένο. Ε, αυτό που προσπαθούμε λοιπόν είναι να αποφύγουμε την ανθρώπινη πλακία. Καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Μπράτπον Λέτε ότι ίσως ε, μπορούν όλα αυτά να τα κάνουμε μέσω των ασφαλιστικών εταιριών, ε, αυτοί που ε, οδηγούν μεθυσμένοι να πληρώνουν πιο υψηλά ασφάλιστρα. Καταλαβαίνω την αρχή, αλλά όπως γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο ακριβή η ασφάλιση που ο κόσμος οδηγεί χωρίς ασφάλιση, το οποίο είναι παράνομο, αλλά προσπαθήστε να τους πιάσετε. Μόνο αν τρακάρουν το αυτοκίνητό σας μπορεί να το ανακαλύψετε αυτό. Και γι' αυτό έχουμε περιπτώσει οπου ε, όπου ε, ε, σκοτώθηκε 16χρονος και ο οδηγός του αυτοκινήτου απλά έφυγε γιατί, διότι ή μεθυσμένος θα ήταν ή δεν θα είχε ασφάλιστη. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπε πολύ σωστά ο, ο κύριος Higgins. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχουμε την πιο καταπληκτική νομοθεσία σε τον κόσμο. Εάν όμως η αστυνομία δεν επιβάλλει τον νόμο, τότε το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και η επίκρισή μου όσον αφορά την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπερβολικά το ότι έχουμε υπερβολικά πολλή νομοθεσία, αλλά το ότι δεν επιβάλλεται ο νόμος ε, από τις αρμόδιες αρχές σε κάποιες από τις χώρες. Ό,τι και να αποφασίσουμε λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να επιβάλλεται ο νόμος και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους διάφορους φορείς, με την αστυνομία για να ε, γνωρίζουμε ότι γίνεται αυτό και επίσης όταν ε, καταλήγει κάποιος στο δικαστήριο δεν αρκεί ένα πρόστιμο 10 ευρώ όταν κάποιος έχει ε, διαπράξει πιο σοβαρό αδίκημα. Ε, δεν είναι λοιπόν το θέμα της επιβολής, είναι και το δικαστικό σύστημα ώστε να διασφαλίσουμε να επιβάλλονται σημαντικές ποινές και γι' αυτό η έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ είναι επίσης σημαντική. Ε, θα πρέπει να μπορούμε να ε, επιβάλλουμε τον νόμο και σε διασυνοριακό επίπεδο, όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων. Ε, πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα προχωρήσει η ψηφοφορία αύριο. Ο κύριος Πασκαρέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελευταία φορά κύριε Πασκαρέλη ή θα έχουμε την... Τελευταία φορά. Εντάξει, τότε θα σας δώσω μόνο δύο λεπτά. Όχι, δεν πειράζει, σας δίνω περισσότερο. Ναι, Πρόεδρε. Θα μπορούσα να αρκεστώ να υπογραμμίσω ότι από την πλευρά της Κομισιόν δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε για το γεγονός ότι η παιδεία και η έλεγχη και οι ποινές είναι το κλειδί για την οδική ασφαλεία. Έχουμε αρκετούς κανόνες, το σημαντικό είναι να τηρηθούν. Θα ήθελα και εγώ να εξε... τη Κομισιόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του σκιώδη εισηγητέ καθώ και όλου όσου παρενέβησαν στη συζήτηση, γιατί όλοι ενισχύουν κατά κάποιο τρόπο το μήνυμα που θέλει να περάσει η Κομισιόν σε αυτέ τι κατευθύνσει γραμμέ για την ε, οδική ασφάλεια που υιοθέτησε πέρυσι και να, υποστηρί... να, στηρί... να υπογραμμίσω κιόλα ότι η κατάσταση στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική διαφοροποιημένοι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιούνις εξελίσσεις ε, από το Αλγάρβε μέχρι τη Λαπονία ή το Τυρόλο. Είναι πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις. Υπάρχει μεγάλος χώρος για την επικουρικότητα, εκπαίδευση, έλεγχη, τήρηση των κανόνων. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αφήσουμε στις εθνικές και ίσως και στις τοπικές αρχές αλλά είναι αλήθεια πως έχει να παίξει ρόλο και η Ευρώπη στον καθορισμό ορισμένων κοινών κανόνων, όπως για παράδειγμα δίπλωμα οδήγησης, ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα αυτοκίνητα, <clears throat> κάποιους κανόνες που αποτελούν το κοινοτικό κεκτημένο. Θα περιοριστώ σε κάποιους ε, προβληματισμούς μόνο για τις συμβιβαστικέ λύσεις. Να πω πρώτα αυτά που αφορούν τον περίφημο συντονιστή της οδικής ασφάλειας, συμβαστική Β. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε, και το συναισθανόμαστε και εμείς στην Κομισιόν, χρειαζόμαστε πιο έντονο συντονισμό ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται ακόμα ένα συντονιστή. Πρέπει να το κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Αυτή είναι μια έκκληση προ την Κομισιόν να οργανωθεί καλύτερα και είναι μια έκκληση την οποία λάβαμε όσον αφορά έναν εξωτερικό πρόσωπο από το Κομισιόν ή από το Κοινοβούλιο για να φέρει το μήνυμα της οδικής ασφάλειας, γιατί όχι, θα μπορούσαμε να αποτελέσει έναν πρέσβη, ας πούμε, καλής βούλησης, όπως αυτή του ΟΗΕ, για τα διάφορα θέματα που έχουν κοινωνική σημασία, γιατί λοιπόν όχι και ένα συντονιστή για την οδική ασφάλεια που θα προσωποποιεί αυτό το ισχυρό μήνυμα της Ευρώπης. Τώρα, όσον αφορά τα εργαλεία βασικά ώστε να ασκήσουμε πολιτική οδικής ασφάλεια. αναφέρομαι στη συμβιβαστική γάμα σε για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Οδικής Ασφάλειας, τροπολογία νη για το σχέδιο Βερόνικα και η τροπολογία σε Έχουμε ήδη ένα παρατηρητήριο για την οδική ασφάλεια στις υπηρεσίες της Κομισιόν. Είναι η βάση δεδομένων μας, είναι το ε, site του ίντερνετ που έχουμε, είναι η μάζα των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε ακόμα ένα κέντρο. Αντίθετα, αν το Κοινοβούλιο στις επόμενες του μέρες ε, μάλλον στις επόμενες συζητήσεις για τα δημοσιονομικά αποφασίσει να μας δώσει και άλλα χρήματα, θα τα εξοδέψουμε καταλήλως. Όσον αφορά το σχέδιο Βερόνικα, το πρόγραμμα Βερόνικα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ακόμα αξιολογούμε τα αποτελέσματά του και θα ήμουν κάπως διστακτικός όσον αφορά την άμεση του εφαρμογή. Θα προτιμούσα να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Τώρα, τροπολογία D, εκπαίδευση, κατάρτιση, υποστηρίζουμε. Αντίθετα, τροπολογία ε, που περιορίστηκε σε διάφορους ομιλητές στο θεζήτημα της εξέτασης της όρασης, που είναι όμως μια ευρύτερη τροπολογία και καλύπτει όλη την επιτυχή των ε, περιοδικών ιατρικών εξετάσεων για τους πιο ηλικιωμένους οδηγούς. Εγώ προσωπικά υποκλίνομαι στα αυτή τη χειρονομία του κύριου Ρίκη και η Κομισιόν να πιστεύει πως δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Να, υπερ... να δηλαδή για πράγματα τα οποία μπορεί να τα εμπνεώμαστε από ανησυχίε που μπορεί να είναι ξέπαινες, αλλά που υπό το φως της επιστήμης δεν είναι βάσιμες. Δηλαδή δεν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ηλικία και την κακή οδική συμπεριφορά και πρέπει να αποφύγουμε και κάθε διάκριση σε σχέση με την ηλικία, με βάση μάλλον την ηλικία. Προχωράμε λοιπόν προς μια συμφωνία για την οδηγία για τις διασυνοριακές διώξεις και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί η Κομισιόν με θέματα ελέγχου ταχύτητας, κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών, χρήση του κινητού τηλεφώνου. Άρα λοιπόν οι τροπολογίες F, Α και Z εμπίπτουν στο πρόγραμμα δράσης που θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας που ελπίζω θα εγκριθεί συντόμως. Όσον αφορά το μετρητή εθιλένης μέσα στο αλκοολόξ, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτέλους για αυτό το θέμα, καταρχήν για να είναι διαλειτουργικά και συμβατά εφηλομετρητέ οι οποίε ε, να είναι αποδεκτοί σε ένα κράτο μέλος, να είναι αποδεκτοί και στα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα τύπο αποδοχή ε, αυτών των μετρητών και για ποιο τύπο οδηγού θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε μέσω μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα ε, ήμουν στο, ε, όμως πιο διστακτικός όσον αφορά την ε, συμβαστική F για την οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή φαρμάκων. Φυσικά και δεν πρέπει κανείς να οδηγεί υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Αλλά και εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απόλυτη και πλήρη απαγόρευση γενική, χωρίς να μελετήσουμε πιο λεπτομεριακά, όπως το κάνουμε με, το, με την έρευνα Druid, ολόκληρη αυτή την προβλήμα, ολόκληρο αυτό το θέμα. Τροπολογία άσο, που ζητά από την Κομισιόν να, να σκεφτεί να ενισχύσει τον έλεγχο και των, των επαγγελματιών οδηγών να τους δώσει ασφαλείς χώρους στάθμευσης κτλ. Αυτά αντιστοιχούν σε αυτό που κάνουμε και σε αυτό που θα κάνουμε με τις κατευθύνες γραμμές για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου. Είναι μια τροπολογία την οποία υποστηρίζουμε, καθώς και αυτή που αφορά τις υποδομές, την, την τροπολογία η GLM επίσης, που αναφέρονται στην ασφάλεια των οχημάτων, τα ΕΦΗ, e, συστήματα μεταφορών. Πρόκειται για θέματα τα οποία εξακολουθούν να είναι μελέτη. Θα δείτε λοιπόν τις εξελίξεις είτε σε νομοθεσίες, νομοθετικά κείμενα είτε σε ανακοινώσεις της Κομισιόν. Οι ευάλωτοι χρήστες τώρα είναι η προτεραιότητα του επόμενου προγράμματος δράσης. Και θα κάνουμε σχετική έκθεση σύντομα για τις διατάξεις είδους ε, καθρέφτη για την νεκρή γωνία κτλ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς είμαστε ευτυχείς που αύριο θα γίνει ψηφοφορία για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοχ. Θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Θέλω. Είναι λίγο περίπλοκο όμως να συνοψίσει κανείς όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση, τη συμφωνία αλλά και για την κριτική. Κοιτάξτε, η έκθεσή μου δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, δεν κάνουμε νομοθεσία. Ενθαρρύνουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παροτρύνουμε και τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες και τους ΟΤΑ να αναλάβουν δράση. Και η κριτική μου δείχνει ότι μερικοί δεν διάβασαν σε λεπτομέρειε το κείμενο. Γιατί σε συγκεκριμένα πράγματα είπαμε, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τώρα με πυροβολείτε επειδή το γράφουμε εδώ, γιατί ζητάμε να το λύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ας το διαβάσουμε και μετά να ψηφίσουμε. Ε, μερικά θέματα ουσιαστικά που επανειλημμένα επικρίθηκαν είναι αυτό η οφθαλμολογική εξέταση. Για τους μεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε υποχρεωτικό, αλλιώς δεν γίνεται. Οι άλλοι λένε ότι ε, το παρακάνουμε. Είναι πολύ διστάμενες οι απόψεις. Δεν θέλω όμως να χαθεί εντελώ το θέμα. Θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι είναι σημαντικό να κοιτάζει τα μάτια του. Και δεν είναι μια, ένας έλεγχος αντανακλαστικών ή κάτι που δεν διορθώνεται ο έλεγχος της όρασης δείχνει ότι αν έχεις πρόβλημα όρασης από σήμερα μέχρι αύριο, από τη μια ώρα στην άλλη μπορείς να τα αλλάξει. Σου βάζουν γυαλιά. Δεν θα σου πάρουν το δίπλωμα. Πρότεινε ο κύριος Βαντάλεν μερικά πράγματα που βεβαίως δεν γίνονται. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν στόχοι, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων στα τροχιά ή των σοβαρά τραυματισμένων, αλλά καλούνται και τα κράτη-μέλη λόγω της ιστορικής τους εξέλιξης, των παραδόσεών τους και τα λοιπά, να κάνουν προγράμματα δράσης. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να επαναπαύονται ότι θα τα ρυθμίσει όλα η Ένωση και συμφωνώ με αυτούς που το είπαν, ε, χρειάζεται κάποιο συντονισμό όμως για να μην τραβάει ο καθένας στο δρόμο του, γιατί έχουμε εσωτερική αγορά, όλοι μετακινούμαστε στους δρόμους της Ένωσης, γι' αυτό χρειάζεται ο συντονισμός, γι' αυτό το ζητάμε. Κύριε Πασκαρέλη. Ακόμα δεν καταλάβατε ότι δεν ζητώ έξτρα συντονιστή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή το είπα εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον. Στο εσωτερικό της Επιτροπής, στις υπηρεσίες της Επιτροπής και ακόμα δεν υπάρχει αυτός ο συντονισμός. Επιμένω, το διατηρώ, όχι καινούριο όργανο. Για τα θέματα του εινοπνεύματος σας είπα, όποιος πιάνει τιμόνι να μην πιάνει ποτήρι. Εγώ δεν μετακινούμαι από αυτό. Ε, Τώρα, αν αρχίσουμε να βάζουμε την κολογγυφιά με τα ποσοστά, εντάξει, μπορεί και κάποιος να πάρει ένα φάρμακο που έχει νόπνευμα ή να πιει λίγο χυμό και να αρχίσει ακολική ζήμωση στο στομάχι του ή μια καραμέλα, δεν ναι, είμαστε υπερβολικοί. Αυτά. Περιμένω με χαρά αύριο την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο κ. Κόκ, λοιπόν, αύριο θα ψηφίσουμε και ελπίζουμε θα περάσει την Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ όλους. Επόμενο θέμα είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τις ε, οδικές παραβάσεις. εξηγήτρια είναι η κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα μας ενημερώσει για τον τριμερή διάλογο που έγινε και σήμερα το πρωί τελευταία. Ξέρω πως σε πέντε ώρα πρέπει να τελειώσουμε, να φύγεις μάλλον. Γι' αυτό σου δίνω μέσο στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγκρατημένη αισιοδοξία νομίζω μπορούμε να πούμε ότι προχωρούμε. Γιατί ξέρετε ότι σε αυτά τα θέματα καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έχω ευχάριστα νέα. Μπορούμε πια να μιλούμε για μια προσυμφωνία, για να μην πω συμφωνία έτσι με κάθε επιφύλαξη και συγκράτηση. Και μιλώ υπό τον έλεγχο των φίλων σχεδόν εισηγητών και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εκείνους και τη γραμματεία και σας προσωπικά πρόεδρε για όλη τη βοήθεια. που μας ε, παρήχαν για να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τη Βελγική Προεδρία, ε, γιατί εκείνη ξεκίνησε Εκείνη δρομολόγησε αυτό το θέμα και ακολούθησε η Ουγγρική Προεδρία και ελπίζω να μπορέσει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας και ε, κάτω από το βλέμμα της. Όπως γνωρίζετε, από την αρχή είχαμε περιορισμούς, είχαμε προβλήματα, ιδίως στο Συμβούλιο υπήρχε ε, μειοψηφία εμπλοκής. Και αν δεν την κερδίζαμε, δεν θα μπορούσαμε ακριβώς να δρομολογήσουμε καθόλου την έκθεση αυτή. Για να έχουν τα κράτη-μέλη μια δυνατότητα στα χέρια τους να μπορούν να επιβάλλουν τις απαραίτητες κυρώσεις και τα πρόστιμα για να σταματήσει αυτή η πληγή των ξένων οδηγών που δεν διέμεναν στη χώρα και δεν ετοιμορούντο. Και αυτό αποθάρρυνε και τις διοκτικές αρχές και την τροχέα γιατί αντιδρούσε ο ντόπιο πληθυσμό, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές ε, ή σε περιοχές με έντονο τουρισμό. Οι μόνιμοι κάτοικοι έβλεπαν τους ξένους και τους τουρίστες κατά το δοκούν να παραβιάζουν ε, τον κώδικα οδικής ε, κυκλοφορίας και να περνούν τα σύνορα και χαίρεται. Να μην τιμωρούνται. Ήταν πολύ δύσκολο να τους εντοπίσει κανείς όσα συστήματα και να έχουμε τηλεματικής. Αν δεν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και επεξεργασία της πληροφορίας εκ των υστέρων, δεν μπορούσε κανείς να τους διώξει πέραν των εθνικών συνόρων του. Πολύ ωραία είπατε κι εσείς προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να ε, διατηρεί και να διευρύνει την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα τη στιγμή που έχουμε ε, διευρυμένη κινητικότητα και αυτό είναι δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών που κινούνται σε όλη την Ένωση. Λοιπόν, ένα πρώτο βήμα έγινε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι και σημαντικό και την ευχαριστώ για τη στήριξή της και την καθημερινή βοήθεια στο θέμα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε ε, ε, δέχτηκαν μια αλλαγή στη νομική βάση για να μπορέσουμε να κινηθούμε και να επιτύχουμε ακριβώς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο στο σύνολό του να συμφωνήσουν και να δεχθούν τις προτάσεις μας για την ανταλλαγή, προχωρήσαμε. Και αν μη τι άλλο, να μην βασιζόμαστε μόνο στην αστυνομική συνεργασία ως ε, νομική βάση, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, να προχωρούμε. Για να μπορέσουμε να εργαστούμε ακριβώς με βάση τη συνεργασία της αστυνομίας μπορεί να είναι περιοριστική από τη μια, από την άλλη μας ανοίγει νέες δυνατότητες. Δηλαδή, έχουμε και τέσσερις επιπλέον παραβάσεις ε, όπου εφαρμόζεται το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και επίσης η δυνατότητα σε μια ε, ρήτρα αναθεώρησης πολύ ισχυρή να λέμε ότι μετά από μια πενταετία, δύο για τη μεταφορά και τρία χρόνια για μια διάμεση έκθεση, να έχουμε κάποια αναφορά, κάποια διαδικαστική αναφορά για την εφαρμογή στην πενταετία. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κάνει μόνο την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτού του πρώτου βήματος, αλλά να κοιτάει τι θα γίνει από εκεί και πέρα και να το διευρύνει σε νέες προτάσεις. Τα κράτη-μέλη είχαν πάρα πολλές επιφυλάξεις για αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, σήμερα δεσμεύτηκε η Ουγγρική Προεδρία να διασκεδάσει και την τελευταία επιφύλαξη. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Και θα πούμε το εξή. Τη στιγμή που αποφασίζει να κινήσει δίωξη η διαδικασία η χώρα στην οποία έχει γίνει παράβαση, θα κινητοποιείται και ε, η χώρα στην οποία είναι καταχωρημένη η πινακίδα του αυτοκινήτου που έχει κάνει την παράβαση. Αυτό πια μπορούμε να το πούμε ε, με βεβαιότητα και ε, να θεωρήσουμε ότι έχει καταλήξει και το ζητούσε το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, είναι ένα από τα σημεία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι συνάδελφοί μου επέμειναν πάρα πολύ γιατί σε αυτό το θέμα που είναι αστυνομική συνεργασία και η χρήση ενός συστήματος ε, πληροφόρησης, αυτό το Ιούκαρις, υπήρχε κάποιος κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα. Τώρα νομίζω ότι αυτός έχει ε, αποσοφηθεί. Το έχουμε λύσει σωστά, δηλαδή όλη η διαδικασία υπόκειται σαφέστατα στην εμπιστευτικότητα στο απόρριτο, στην προστασία, στη δυνατότητα να πάσα στιγμή ο ενδιαφερόμενος να απαιτήσει και από τα δύο κράτη το δικό του και εκεί που έγινε η παράβαση ε, να απαιτήσει λέω να του δώσουν τα στοιχεία που αντίλεξαν για να τα γνωρίζει κτλ. και να γίνεται ε, αποκλειστική χρήση ακριβώς για αυτό το λόγο που ε, χρειάζονται τα στοιχεία και για τίποτα άλλο. Αυτό τουλάχιστον το κλειδώσαμε. Στις κατεξουσιοδότηση πράξης, επίσης ήταν πολύ ισχυρή αντίσταση από πλευράς κρατών μελών, γιατί και στο κεφάλαιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφώνησε, το έχει ζητήσει, για την τεχνική προσαρμογή ε, του παραρτήματος 1 για την πιο αυτόματη εφαρμογή αυτού του συστήματος. Θέλαμε όχι μόνο να μπορεί να εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους δύο κανόνες αστυνομικής συνεργασίας, αλλά και αλλού. Να μπορέσει να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτού του παραρτήματος που αναφέρεται στις 8 παραβάσεις, στην προστασία δεδομένων, ε, στην ανταλλαγή προφοριών. Εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ τεχνικά, δεν θέλω να σας κουράσω. Ε, μετά την πενταετία να ε, βελτιώνεται αυτό. Μέχρι τώρα το Συμβούλιο είχε πολύ ισχυρέ επιφυλάξεις δεν ήθελε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα και το δεχόμενο γιατί ε, υπερεύαινε κατά πολύ την αστυνομική συνεργασία. Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση και χάρη στην επιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, στην πυγμή της Ουγγρικής Προεδρίας νομίζω ότι θα ανακτήσουμε τη δυνατότητα και οι κατεξουσιοδότηση πράξεις να λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την νομοθεσία και όχι μόνο την αστυνομική συνεργασία. Η ευθύνη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κύριο Βαντάλεν. Το καταφέραμε, γιατί τι μα είχε ζητήσει ο κύριο Βαντάλεν. Και ο κύριο Κράμερ, νομίζω, και ο κύριο Μπαχ. Να διευκρινίσουμε τη νομική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εξήγησε ότι αυτές οι δηλώσεις που δεν είναι αμυγός πολιτικές ε, προκαλούσαν κάποιο πρόβλημα για να τις δώσουν γραπτός. Γιατί λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ε, στο πεδίο ε, ταυτοποίησης της ευθύνης την κρατική νομοθεσία. Χωρίς αυτό να αντιφάσκει με την νομοθεσία του άλλου κράτους. Όπως γνωρίζετε κύριε Φατάλε και οι άλλοι συνάδελφοι όλοι αντέδρεσαν πάρα πολύ κάποια κράτη η Γερμανία, γιατί έχει πολύ ρητές ρυθμίσεις περί και το λέει και με ξεχωριστή δήλωση στην κοινή θέση. Εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σημείο που μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξηγήσει καλά, με σωστό τρόπο, αυτό μας πρότειναν και τους πιστεύουμε, το είπε και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής σήμερα και με γραπτό τρόπο. Και να είναι λίγο πιο ευρία η διατύπωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί μόνο να βάλει χειροπέδες στα ε, ε, ίδια της στα χέρια να μην μπορεί να δράσει και να διακυβευθεί όλη η συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, η Κομισιόν δεσμεύεται να ε, κάνει μια διατύπωση γραπτή, μεν πλην όμως λίγο πιο χαλαρή και όχι τόσο αυστηρή για την εφαρμογή, για να μπορέσει να εφαρμοστεί και στην Ολλανδία. Αλλιώς, στην Ολομέλεια μπορεί να κάνουν μια ανακοίνωση πιο στεναρή, ας πούμε, ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Κάλλας και να γραφτεί στα πρακτικά του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ακόμα ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και ε, η διατύπωση ε, αυτή θα έρθει, μας το διαβεβαιώνει και η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη γραπτή εκδοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν μας καλύπτει αυτό, δεν μας ικανοποιεί, να έρθει να τα πει στην Ολομέλεια ο Αντιπρόεδρος κύριος Κάλλας, ρητά λόγια ράτα που να μείνουν στα πρακτικά του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Ρικέ ανησύχησε για το, τη συστημένη επιστολή. Αυτό είναι τη λογική σκέψη προς το παρόν. Αλλά μας ενδιαφέρει. Δεν είναι και κανένα τρομερό, κανένα τραγικό ζήτημα. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο κύριος Ρικέ. Αλλά αν είχαμε πετύχει όλα αυτά που ζητούσαμε στην πρώτη ανάγνωση, εγώ με μεγάλη μου χαρά θα δεχόμουν και το συστημένο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει για τα βασικά θέματα. Και θα παρακαλούσα κύριε Ρικέ να το δεχτούμε, γιατί το έχουμε συζητήσει και όλοι οι σκιώδες, στην αιτιολογική σκέψη που μόλις αναγνώρισε το Συμβούλιο την ανάγκη να διατηρηθεί αυτό Δηλαδή να παίρνει την επιστολή μόνο ο ενδιαφερόμενος εμπιστευτικά. Αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι θα το λαμβάνει. Αλλά αυτό δεν είναι ε, διαδεδομένη πρακτική στα κράτη-μέλη, ούτε για τους πολίτες τους. Δεν τους έλουν συστημένο γράμμα για μια παράβαση, για να βεβαιώσουν το πρόστιμο. Ούτε καν στη Γαλλία δεν γίνεται αυτό. Οπότε το βάλαμε στην αιτιολογική σκέψη για να συζητηθεί. Επίσης σας ζητώ να με υποστηρίξετε και οι συντονιστές και οι υπόλοιποι για την κοινή δήλωση που προτείνει και το Συμβούλιο. Κάνουμε κοινή δήλωση με το Συμβούλιο. 27 κράτη-μέλη υπέρ της ε, συζήτηση για τους πίνακες ε, συσχετισμών Αυτό που συμφωνήσαμε για την Ευρωβινιέτα, ας πούμε, δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για να προχωρήσουμε. Έχει περίπου κλείσει ε, αυτό το θέμα της έκθεσής μου σε όλα τα στιγμή, εκτός από τους πίνακες αυτούς. Μας ε, προσφέρει τη δυνατότητα το Συμβούλιο να προχωρήσουμε με κοινή δήλωση και νομίζω ότι ε, καλό θα ήταν να πείσουμε και το Κοινοβούλιο ότι είναι πολύ καλή συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπακ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ε, να συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια της ε, κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Ε, πιστεύω ότι έχει βρεθεί πολύ καλό συμβασμός εδώ πέρα να... Ευχαριστήσω και την Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία διότι είχε μπλοκάρει πριν ε, κάνα δύο χρόνια το συγκεκριμένο θέμα και μπόρεσε να προχωρήσει μόνο με την ε, τροποποίηση της ε, νομικής βάσης. Αυτό οδήγησε σε κάποιες δυσκολίες οι οποίες αναφέρθηκαν. Η τροποποίηση της νομικής βάσης μας έχει δώσει κάποιες δυνατότητες όπως την διεύνηση των ποινικών μέτρων. Μας έχει φέρει όμως και κάποιες δυσκολίες διότι τώρα απαιτείται ομοφωνία από το Συμβούλιο, κάτι που έχει οδηγήσει σε σημαντικές δυσκολίες. Ε, όπως επίσης και η διαφορετική νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη που πάντα οδηγεί ε, σε συζητήσεις. Πολύ σύντομα κάποιες παρατηρήσεις. Ε, πιστεύω ότι ε, ελάχιστοι από εμά είναι νομικοί και γι' αυτό Επανελειμμένα χρειάστηκε να συνοηθούμε με την νομική υπηρεσία. Ε, ωστόσο, ε, απαιτείται εμπιστοσύνη από την πλευρά μας και όπως υπόθηκε από την αρχή, πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα συμβιβασμό ο οποίος μας έχει φέρει πολύ κοντά στο στόχο και πρέπει να το στηρίξουμε. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη νέα πρόταση. Η υποχρέωση ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτή από εμά. Το θέμα της ευθύνη. Ε, και τις ε, εγγύσεις για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Πιστεύω ότι στο θέμα αυτό η Κομισιόν έχει συνεργαστεί καλά με την Προεδρία και μπορούμε να στηρίξουμε το θέμα αυτό όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ε, είμαστε κάπως απογοητευμένοι. Το Κοινοβούλιο είχε εδώ μεγαλύτερες φιλοδοξίες, περισσότερες επιθυμίες, οι οποίες όμως ε, στο πακέτο για τα δεδομένα ε, διασφαλίζεται και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε και την πρόταση υπό την παρούσα μορφή. Πιστεύω ότι έτσι έχω συμφωνήσει ως προς τα θέματα που μας ενδιαφέραν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα 7 ομιλητές και λιγότερα από 15 λεπτά για αυτούς και για την Κομισιόν. Παρακαλώ λοιπόν να είσαστε σύντομοι και να σας καλέσω να μην επαναλαμβάνετε όλα όσα ήδη έχουν υποθεί. Καταλαβαίνω ότι υπόθηκαν όλα, όχι όμως από όλους. Σας παρακαλώ βοηθήστε με όμως εδώ πέρα, διότι πρέπει να κλείσουμε στις 5 η ώρα. Η κυρία Σαβισάρ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιάλα Σέντερ ε, και ε, τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ε, ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. χαίρομαι που καταλήξαμε σε συμφωνία ικανοποιητική έχουμε καταλήξει σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. σε καλή συμφωνία με την ε, Επιτροπή. Ε, υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία δεν με ικανοποιούν. Πρώτον, το γεγονός ότι Ε, τα διασυνοριακά δικήματα δεν ε, θα ε, διώκονται μόνο με την ανταλλαγή πληροφοριών. Μετά από πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή. Δεν μπορούσαμε όμως να συμπεριλάβουμε εδώ την δυνατότητα η Κομισιόν να υποβάλει νέες προτάσεις. Έχουμε αναφερθεί στην ανταλλαγή δεδομένων. αλλά η ανταλλαγή δεδομένων υπό τη μορφή που συζητήσαμε σήμερα το πρωί δεν θα είναι ικανοποιητική. Τα κράτη-μέλη στον οποίο το έδαφος ε, έχει πραγματοποιηθεί ε, ε, μια ποινική ενέργεια δεν Ε, θα γνωρίζουν αν ε, οι πληροφορίες έχουν φτάσει στον, σε αυτόν που διέπραξε ε, το αδίκημα, διότι σε κάποια δεν υπάρχουν πλήρη μητρώα κατοικίας. Δεν είμαι επίσης ικανοποιημένη με το γεγονός ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει πίνακες αντιστοιχίας στο διατακτικό του κειμένου. Αναφερόμαστε απλά τους ισχύοντες κανονισμούς ε, στα εκτιμώντας. Και επίσης δεν μ' αρέσει το γεγονός ε, ότι ε, δεν είναι νομοθετική έκθεση αυτή. Αυτό βρίσκω ότι είναι πολύ σοβαρό. Δεν θέλω όμως να επικεντρωθώ στα αρνητικά μόνο. Έχουμε σημειώσει πρόοδο και ελπίζω ότι θα γίνουν πιο ασφαλείς οι ευρωπαϊκοί δρόμοι με την υιοθέτηση του κειμένου αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρο κύριος Βαντάλεν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ένα θέμα θέλω να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ερμηνεύσει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Και εννοώ αυτό που έκανα τροπολογία με τον κύριο Μπαχ πώς ε, θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ευθύνης του οδηγού. Θα παρακαλούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το γράψει αυτό και έχουμε ακούσει πολλά προφορικά, αλλά θέλω γραπτή δήλωση. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το ερμηνεύει και για την ομάδα μου είναι και ζήτημα κομβικό για το εάν θα το αποφασίσουμε ή όχι. Ε, ε, θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ακριβώς βρισκόμαστε εκεί. Λίχτεμπεργε. Äh, ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Γιάλα Σέντερ που κατάφερε από αυτή την πολιτική εμπλοκή του Συμβουλίου τουλάχιστον να κινήσει λίγα πράγματα και να ε, μοιάζει αυτό που μας έφερε με αυτό που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Μιλούσαμε για την οδηγία αυτή για την ποινική ε, δίωξη στην αρχή, τη διασυνοριακή και καταλήξαμε να μιλάμε για διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών. Και το θέμα της αλλαγής της νομικής βάσης δείχνει ότι είναι μάλλον περιθωριακό το θέμα της δίωξης. Αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη είναι να συλλέγουν ε, στοιχεία και δεδομένα. Είναι πρόθυμα να το κάνουν αυτό. Ε, χωρίς προστατευτικές διατάξεις. που κανονικά ε, θα έπρεπε να ισχύουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό έχω κάποια προβλήματα τώρα. Στο μεταξύ δεν έχουμε καταλήξει στην ομάδα μας εάν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Γιατί όλο αυτό το θέμα της προστασίας των δεδομένων έχει παραγωνιστεί και έχει μπει σε αιτιολογικές σκέψεις και δεν είναι στο διατακτικό. Μα ε, αυτό τελικά είναι σύσταση, δηλαδή μια τρύπα στο νερό για την εφαρμογή. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή μέχρι εκεί μας έσυρε το Συμβούλιο και μετά από τεράστια πίεση. Να συλλέγουν στοιχεία δηλαδή, ατάκτως ερημένα και κατά το δοκούν, ε, αλλά χωρίς να βγάζουν τις απαραίτητες ε, συνέπειες, τα απαραίτητα συμπεράσματα και ούτε να ευθύνεται κανείς. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποια κράτη-μέλη. Δεν έχει λυθεί. Ακόμα το συζητούμε. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από το Συμβούλιο που αποδυνάμωσε τόσο πολύ το σημείο και για τους πίνακες αντιστοιχίας αυτό το περιμένουμε πάντα από το Συμβούλιο. Και όταν δεν έχουν κανένα επιχείρημα να αρνηθούν πρόταση του Κοινοβουλίου, αρπάζονται από αυτούς τους πίνακες και ε, νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε να έχουμε πεταριώδη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Κύριε Γκρός, ε, είστε σύντομος, θα σας ήμουν ευγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στη, ε, στη σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση αυτή και την έκθεση ΚΟΧ. Και να σας θυμίσω ότι είναι πολύ κρίμα, αποτελεί σχεδόν ηρωνία ε, το ότι ε, καταβάλουμε προσπάθειες για την ε, οδική ασφάλεια από τη μία, ε, από την άλλη ότι ε, μας εμποδίζουν όσον αφορά την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΛΚ θα στηρίξει το συμβασμό όσο μικρό και να είναι το βήμα αυτό. Είναι μικρό όμως και το Συμβούλιο θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι αν αύριο η προστασία των δεδομένων γίνει πιο σημαντική αύριο από την προστασία των ανθρώπων, τότε αυτό είναι λάθος. Και επίσης, Ε, εάν δημιουργήσουμε εδώ πέρα εμπόδια, αυτό θα εξυπηρετήσει μόνο τους ανθρώπους ε, οι οποίοι ε, οδηγούν με μία ασφαλή τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς ως κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσουμε να ξεμπλοκάρει το θέμα. Για το μπλοκάρουν οι υπουργοί στα διάφορα συμβούλια. Νομίζω ότι μου φαίνεται ότι δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι άνθρωποι τώρα πια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ε, θα είμαι πολύ σύντομη προς χαρά του Προέδρου όσον αφορά ε, την προστασία των δεδομένων. Συμφωνώ με την κυρία Λίχτενπεργκερ. Δεν έχει... Ε, αναφερθεί επαρκώς στο θέμα, η προστασία των δεδομένων και η προστασία των ε, ανθρώπων. Και όσον αφορά την ε, ευθύνη, συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Η κυρία Τίκα. Δεν υπάρχει εμβολία, Όπω ήδη υπάρχουν ε, διμερεί συμφωνίε ανάμεσα σε γειτονικέ χώρε σε σχέση με τη διασυνοριακή επιβολή. Αυτό αποδεικνύει ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε μια οδηγία που καλύπτει το θέμα. Να τονίσω επίσης πως η οδηγία αναφέρεται μόνο στις ε, οικονομικές ε, κυρώσεις, ε, δεν μιλά για ακύρωση του διπλώματος ή αναστολή ισχύω του κτλ. Και αυτά όλα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι όσον αφορά τον δράστη της παραβίασης θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το καθεστώ των περιορισμών γιατί διαφορετικές νομοθεσίες έχουν, έχει κάθε χώρα. Επίσης θέλω να αναφέρω πως διάφορες χώρες φέρουν το κόστος για τη συντήρηση του λογισμικού που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4. Πιστεύω πως και αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ωστόσο την κυρία Γιαλασάνδρη για την εξαιρετική έκθεση. Ελπίζω πως η οδηγία θα είναι πολύ ε, ισχυρή. Έχουμε η χώρα σας και η χώρα μας δεν έχουμε αυτόματα ε, αστυνομική συνεργασία. Όταν συζητήθηκε το θέμα στις 2 και 3 Μαρτίου δεν είχαμε κυβέρνηση, στο Συμβούλιο θέλω να πω, αλλά θα περάσει από το Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε καινούργια κυβέρνηση και πιθανότατα θα υιοθετηθεί. Και έτσι ερχόμαστε στο δικό μου ερώτημα, γιατί σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω πως η κυρία Γιάλα Σέντρη και ο Σκιώδης εισηγητής έκαναν ε, εξαιρετική δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες και σας συγχαίρω. Αλλά Άλλη μια φορά τα ίδια, όπως είπε και ο κύριος Γκρός, ότι οι διάφορες χώρες βγάζουν απ' έξω την ουρά τους. Γιατί επιτρέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο σε τέτοιες υποθέσεις. Ε, άμα θες να είσαι Ευρωπαίος, να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία και ευρωπαϊκή προοπτική για τα θέματα, Όπου πρόκειται για διασυνοριακή ανταλλαγή. Γιατί επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να απουσιάζουν. Και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν. δεν έχει νόημα. Ακόμα και ένα κράτος να κάνει opt-out, να μείνει απ' έξω, πραγματικά το θεωρώ αναησία. Απελπίζομαι με την ίδια μου τη χώρα, αλλά εντάξει δεν είναι και τίποτα καινούργιο αυτό. Ο κύριος Ρόιτερ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι καταρχήν Συμμερίζομαι τη δική σας ανάλυση. Να ευχαριστήσω ωστόσο την, καταρχήν την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές που προσπάθησαν να σώσουν ό,τι γινόταν να σωθεί σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Γνωρίζετε ότι κάναμε αρχικά πια στη νομική βάση και ε, είχαμε μάλιστα αποκλείσει τη δυνατότητα του opt-out. Σε κάποια φάση όμως συνειδητοποιήσαμε πως δεν υπήρχε περίπτωση να υιοθετηθεί αυτή η οδηγία από το Συμβούλιο επί τη βάση αυτής της νομικής βάσης. Και έπειτα ελιχθήκαμε, εμείς ήμασταν σε πολύ δύσκολη θέση και ε, θεωρήσαμε πως η νομική βάση θα έπρεπε να είναι η νομική βάση για τις μεταφορές και άρα το Συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει με ομοφωνία. Θα πρέπει να πω λοιπόν ότι επί τη βάση της δυσκολίας αυτών των διαπραγματεύσεων είμαι ευτυχής που καταφέραμε έστω και αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Ξέρετε ότι μετά από πέντε χρόνια θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεταρρύθμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να σας πω όλα τα στοιχεία. Υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές, ε, ουσιαστική προστασία του πολίτη στο άρθρο 7 της οδηγίας, όχι μόνο στα εκτιμώντας, αλλά και στο άρθρο 7 Υπάρχει ένα ενημερωτικό, μια ενημερωτική επιστολή με τρι, μια διαδικασία τριών φάσεων. Αυτό το, αυτή η επιστολή θα μεταφραστεί ήδη στην οδηγία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ακόμα και αν δεν είναι υποχρεωτικό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, και σε σχέση με τις άλλες οδηγίες, τις σχετικές, όπως ας πούμε η τελευταία για την Ευρωβινιέτα που είχαμε, ε, να απαντήσω όμως Στον κύριο Βαντάλαν είπατε πως ε, ήσασταν πρόθυμος σε μια γραπτή δήλωση να επιβεβαιώσετε ότι ο αντιπρόεδρος Κάλλας ε, διαβάζει την πρόταση οδηγίας, ερμηνεύει μάλλον την πρόταση οδηγίας με τον εξή τρόπο, ότι εφαρμογή δηλαδή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια των δρόμων σημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος ε, που έχει γίνει παραβίαση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει για να διαπιστώσει ποιος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη παραβίαση ε, παρα, άσχετα από την νομοθεσία που ισχύει σε άλλα κρατημέλη. Ακριβώ αυτή την ερώτηση θέσατε κι εσείς. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την Θα πρέπει να ελέγξω αν μπορώ να σας στείλω αυτή τη διατύπωση. Κάθε άτομο έχει προσωπική ευθύνη, αλλά και κάθε κράτος μέλος. Αυτό αφηνίζεται και πιστεύω πως με αυτά τα στοιχεία, Πρόεδρε, θα έχετε αρκετά στη διάθεσή σας, ώστε να ολοκληρώσετε τις συζητήσεις σας και ελπίζω πως το τέλος θα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο γιατί κάποια στιγμή πιστεύαμε πως αυτή η νομική πρόταση είχε αποβιώσει και δεν θα προχωρούσε καθόλου. Μας βοήθησε η Βελγική Προεδρία, η Ουγγρική Προεδρία και το Κοινοβούλιο και σώσαμε ό,τι γινόταν ακόμα να περισωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ρόιτερ, κυρία Γιαλασέντερ. Κυρία Γιαλασέντερ κινδύνευσε να είναι η πιο μακρά εισηγήτρια στην ιστορία αυτής της Επιτροπής. Το πρώτο βέβαια ρεκόρ το έχω εγώ για την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Και ευτυχώς θα παραμείνω κάτοχος του ρεκόρ. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι κατάλαβα θα περάσει από την Ολομέλεια τον Ιούλιο και ευχαριστώ την εισηγήτρια και όπως είπα και τους και εισηγητές για τη σκληρή δουλειά και την Επιτροπή. Μπράβο σε όλους. Σύντομα, ένα λεπτό γιατί έχουμε τους συντονιστές και μετά έχω και μια ανακοίνωση πριν φύγετε όλοι. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταλαβαίνω τώρα ε, τη στάση σας κα, καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης. Δεν θέλετε να χάσετε το ρεκόρ σας. Τώρα το πιάσα. Δεν πειράζει. Με χαρά σας το παραχωρώ, δεν θέλω να το σπάσω. Για το άρθρο 7, για την προστασία των δεδομένων, έχει ενισχυθεί. Είχε γίνει μια, αναφορά στην κοινή θέση για το ΠΡΟΥΜ. Ε, τώρα είναι πραγματικό <coughs> σημείο με τρεις παραγράφους που ανταποκρίνεται πραγματικά σε όλα τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Όλο το άρθρο 7 έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα για να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Δέχτηκαν δε και τις τροπολογίες μας. Παρακαλώ και την κυρία Λίχτεμπερ και την κυρία Μάης να το ξαναδιαβάσετε. Για το opt-out που είπατε ισχύει, αλλά κάτι που έκανε η Ουγγρική Προεδρία είναι το εξή. Στο τεχνικό παράρτημα που εφαρμόζεται το σύστημα ανταλλαγή απόψεων, κατάφερα και συγχαίρω γι' αυτό την Ουγγρική Προεδρία να μπορεί να εφαρμόζεται στα τρία κράτη που έχουν opt-out στη νομική βάση. Δηλαδή το διατηρούν, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό το Ιούκαρι. Και για τους πίνακες αντιστοίχησης παρακαλώ την κατανόηση των συναδέλφων που του ζητούν. Καταφέραμε τουλάχιστον τα 27 κρατημέλη να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να καθίσουν να δεχτούν αυτούς τους πίνακες. Στο άρθρο 10, σημείο 2 και στην αιτιολογική σκέψη 17 γίνεται λόγος για πρώτερη αναγνώριση, αλλά η κοινή δήλωση, η ανακοίνωση μας αρκεί ως κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Πριν συμφύγετε, θέλω να σας πω το εξή. και ο Χάνε, που ήταν στη γραμματεία για μα ε, μια τετραετία, συμμετέχουν για τελευταία φορά στι εργασίε μα. Θα πάνε τώρα στι προκλήσει τη Επιτροπή Βιομηχανία. Ήτρε, καλή δύναμη. Και είμαι βέβαιος ότι δεν συγκρίνεται η Ήτρε με τη δική μας Επιτροπή, αλλά ε, πιστεύω ότι θα διαπρέψετε και εκεί. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων για τα τελευταία χρόνια, τα τέσσερα χρόνια που συνεργαστήκαμε. Mr. Και αφού έφυγε ο κύριος Πασκαρέλη, έφυγε κύριε Ρόιτερ, έτσι Έφυγε. Όχι. Σε δέκα μέρες φεύγει. Εγώ ρώτησα αν έφυγε από την Επιτροπή μας, γιατί ήταν εδώ προηγουμένως. Παρακαλώ να του ευχηθείτε τα καλύτερα για τη σύνταξη. Βλέποντας τα πράγματα όπως πάνε στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σοφό που παίρνει τώρα σύνταξη. Αλλιώ μπορεί να φτάνει και 110 πριν συμπληρώσει ηλικία συνταξιοδότηση, αν δούμε τι κάνουν οι κυβερνήσει μας. Λοιπόν, να το διαβιβάσετε τις θερμότερε ευχές παρακαλώ τη Επιτροπής μας για την αφιπηρέτησή του. Μάλιστα, κύριε Ρόιτερ, θα το πράξω. Καλώς, ακολουθούν συντονιστές σε 5 λεπτά. Μια σύντομη διακοπή και ξαναρχόμαστε.